So, uh, Συνάδελφοι, πάμε στο σημείο 11 της ατζέντα της ΕΚΟΝ. Ανταλλαγή απόψεων με την ε, Κότσεβα, κυρία Κότσεβα, ε, Γενική Διευθύντρια της ε, Eurostat. Uh, Καλωσορίζω, καλώς ήρθατε. Είναι η πρώτη σας φορά που εμφανίζεστε εδώ ως Γενική Διευθύντρια της Eurostat. Διοριστήκατε την 1η Μαρτίου. Πριν είσαστε, ασκούσα τα καθήκοντα της Γενικής Διευθύντριας και έχουμε μια καλή συνεργασία ήδη. Σας συγχαίρω για το διορισμό σας και περιμένω να συνεχίσουμε αυτή την εποφελή συνεργασία σε διάφορους τομείς που συμπεριλαμβάνουν τους νομοθετικούς φακέλους, που είναι, είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε ήδη σε τριμερείς διαλόγους. Σας δίνω πάρα αυτό το λόγο για να κάνετε μια εισαγωγική δήλωση και συνεχεία οι συνάδελφοί μας θα σας υποβάλουν κάποια ερωτήματα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα σας. Όσοι είσαστε σε αυτή την αίθουσα, ξέρετε ότι οι στατιστικές βοηθούν τις επιχειρήσεις, τους πολιτικές και, και εσάς να παίρνετε σημαντικές αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών. Οι στατιστικές είναι σημαντικές και για τους δημοσιογράφους που εξηγούν τις αποφάσεις στο κοινό και εξηγούν και τα νούμερα. Οι στατιστικές έχουν σημασία, όλο και περισσότερη σημασία, για τους Ευρωπαίους πολίτες που θέλουν να παίρνουν αποφάσεις με τα λόγου γνώσεως στην ιδιωτική του ζωή, αλλά βοηθούν και τους πολίτες να διαφοροποιούν ανάμεσα στους πραγματικούς αριθμούς και στα fake news. Όλοι πιστεύουμε λοιπόν ότι οι στατιστικές έχουν σημασία. Και επειδή έχουν σημασία, κυρίες και κύριοι, φανταστείτε πόσο προνομιούχα αισθάνομαι και πόση τιμή αισθάνομαι που με διόρισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως τη νέα Γενική Διευθύντρια και θα είμαι στο τιμόνι των δύσκολων αυτών καιρών στη Eurostat. Σας ευχαριστώ που λίγο καιρό μετά το διορισμό μου μου δώσατε δυνατότητα να έρθω εδώ για να σας παρουσιάσω τις απόψεις μου, τις προτεραιότητες της στατιστικής μας υπηρεσίας τα επόμενα χρόνια. Θα ήθελα πάρα αυτά. Παρότι είπε ο κ. Γκουαλτιέρη ότι ήμουνα ασκούσα τα καθήκοντα της Γενικής Διευθύντριας για πάνω από ένα χρόνο και είχαμε τακτικές επαφές, να σας πω ότι δεν θα είναι η σημερινή η τελευταία μου εμφάνιση εδώ και η συνεργασία μου μαζί σας δεν θα περιορίζεται στον ετήσιο στατιστικό διάλογο που προβλέπετε και νόμου. Αυτό γιατί πιστεύω στεναρά, αν μου επιτρέπετε τις συγκρίσεις, ότι υπάρχει κάτι κοινό ανάμεσα στα δύο θεσμικά μας όργανα κυρίως, ότι τροποντινά τα δύο μας όργανα παίζουν σημαντικό ρόλο ούτω ώστε να προωθήσουμε τη δημοκρατία, τη διαφάνεια και την ε, λογοδοσία των ε, δημοσίων φορέων και της πολιτικής. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε αυτό το μόνιμο διάλογο εμείς η Στατιστική Υπηρεσία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να είναι ανοιχτός ε, αυτός ο διάλογος και αποτελεσματικός. Γι' αυτό λοιπόν, Πρόεδρε και αξιότιμοι βουλευτέ, να σα πω ποιε είναι οι ιδέε μου για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι ευρωπαϊκέ στατιστικέ. Όλοι συμφωνούμε ότι έχουν σημασία οι στατιστικέ και βλέπουμε παντού ότι οι στατιστικέ είναι εκ των όνου κάνευ για τι αποφάσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση και για την μέτρηση των επιδόσεων και την επίπτωση διαφόρων ευρωπαϊκών πρωτοβουλειών και δραστηριοτήτων. Υπάρχουν πάρα πολλά ε, παραδείγματα ε, υψηλά, υψηλής ποιότητας ε, νούμερα σορευτικά νούμερα υποστηρίζουν το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη, ε, το σχέδιο ε, σταθερότητα και ανάπτυξη, την οικονομική διακυβέρνηση, του στόχου τη βιώσιμη ανάπτυξη, το ευρωπαϊκό εξάμεινο και. Α βάλω μια τελεία εδώ, γιατί θα μπορούσα να τελειώσω, ε, να συνεχίσω ατέρμονα. Παράλληλα, σκεφτόμουν σήμερα πώς να σας παρουσιάσω τις ιδέες μου για το μέλλον. Δεν μπορώ να σας παρουσιάσω τις συγκεκριμένες προτεραιότητες χωρίς να σας περιγράψω εν συντομία ποια είναι η πραγματικότητα μέσα στην οποία ε, ετοιμάζονται οι ευρωπαϊκές στατιστικές. Αυτή την ε, πραγματικότητα την αντιμετωπίζουν όλοι οι πολίτες αυτόν τον εξελισσόμενο χρόνο και διαμορφώνονται από δύο τάσεις. Ε, γρήγορη εξέλιξη της ψηφιακής τεχνολογίας ή τεχνολογιών και η έκρηξη των πληροφοριών. Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιου τύπου πράγματα ποτέ στο παρελθόν. Σήμερα οι Ευρωπαίοι πολίτες ε, είναι ψηφιακά ενήμεροι, είναι καλωδιο... καλωδιωμένοι με παγκόσμιο τρόπο και έχουν πρόσβαση σε νούμερα. Οι επίσημες στατιστικές ε, δεν είναι μόνο νούμερα, αυξάνουν τον αριθμό παρόχων ε, αριθμών άλλων από άλλες πηγές μη επίσημες ε, που ανταγωνίζονται σε επίσημες. Για μας λοιπόν, για τις, ε, τους επίσημους στατιστικολόγους, αυτό είναι μια πρόκληση. Μια πρόκληση. Καταρχάς να έχουμε σημασία, δεύτερον να είμαστε γρήγοροι και τρίτον να είμαστε μια αξιόπιστη πηγή. Γιατί δεν ε, έχουμε πλέον το μονοπόλιο που είχαμε πριν από κάποια χρόνια ότι είμαστε, που ήμασταν η μόνη πηγή ενημέρωσης. Επομένως, με αυτές τις ε, προκλήσεις στο μυαλό είμαι πεπισμένη ότι η εποχή που αυξάνουν τα στατιστικά νούμερα και χρησιμοποιούνται και για διαμόρφωση πολιτική και για πολιτικούς σκοπούς και για διαμόρφωση προεκλογικών ε, ε, στρατιών, να έχουμε ας πούμε αξιόπιστα στοιχεία είναι απαραίτητη. Είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που θα ήθελα να σας, αντιμετωπίσω. Αυτό είναι το όνειρό μου. Όταν ας πούμε ταξιδεύεις κάπου και μιλάς ας πούμε ε, με τον ταξιτζή για διάφορα θέματα, για το πληθωρισμό, για τη μετανάστευση. Και χωρίς να ξέρει ο ταξιτζής ε, που δουλεύω, ο ένας ταξιτζής μια φορά μου είπε πήγαινε στο, στη στην ιστοσελίδα της Eurostat να δεις εκεί τα νούμερα. Αυτό θα ήταν ένα όνειρο να συμβεί βέβαια. Ελπίζω κάποια στιγμή να υλοποιηθεί. Ε, και επειδή για πρώτη φορά έρχομαι ενώπιόν σας, θα ήθελα να σας πω κάποια απλά στοιχεία από την καριέρα μου. Ε, στην επαγγελματική μου καριέρα ξεκίνησα στον ακαδημαϊκό χώρο. Αυτή ήταν πολύ σημαντική περίοδος ε, που μου έδωσε μια φυσική περιέργεια να βρίσκω εφάνταστες λύσεις σε συχνά δύσκολα προβλήματα. Ε, συνεχεία, μετά τον ε, πανεπιστημιακό χώρο ε, ήμουν επικεφαλής ε, της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, που ήταν πολύ επιτυχής περίοδο, γιατί απέκτησα εμπειρία και κατάλαβα πόσο σημαντικά είναι τα νούμερα. Πρέπει να είναι αντικειμενικά, να είναι έτοιμα γρήγορα, να είναι αντικειμενικά για να παίρνω τις σωστές πολιτικές. Και τα τελευταία έξι χρόνια ήμουνα σε υψηλές θέσεις στη Eurostar. Ε, καταρχάς ήμουν αναπληρώτρια γενική διευθύντρια και όπως είπε και ο πρόεδρο. Ε, για πάνω από ένα χρόνο ε, ασκούσα τα καθήκον της Γενικής Διευθύντριας και αυτό μου έδωσε μια πανευρωπαϊκή εμπειρία και προοπτική. Αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι όλες αυτές τις διάφορες εμπειρίες να τις ε, συγχωνεύσω για να αντιμετωπίσω τις σημερινές προκλήσεις. Τώρα θα ήθελα να σταθώ σε τρεις σημαντικές προτεραιότητες που συνοψίζουν και τις προθέσεις που ε, θα, θα δείτε ότι έχω τα επόμενα χρόνια. Κα, καταρχάς, η εστίασή μου θα αφορά την παραγωγή στατιστικών. Μπορεί να θεωρείτε ότι αυτό είναι τετριμένο, ότι είναι ούτως ή άλλως αρμοδιότητα της Eurostar. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε μια επικριτική αναθεώρηση. Ε, που έχουν σημασία οι στατιστικές που παράγουμε, είναι καλές ε, με, βάση τις ανάγκες και που ε, δεν είναι αρκετά γρήγορες αν βλέπω, αν ε, θέλω να εστιάσω στο πού πρέπει να ε, δώσουμε μεγαλύτερη σημασία και να είμαστε καλύτεροι, είναι να είμαστε πιο γρήγοροι, ειδικά στις, ε, κοινωνικές, στις στατιστικές για κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα. Μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή πολλά από τα ευρωπαϊκά οικοδομήματα είναι υπό εξέταση, πολλές μεταρρυθμίσεις είναι εξελίξη και όλα αυτά απαιτούν ε, αναθεώρηση με κριτικό μάτι των ευρωπαϊκών στατιστικών. Μερικά παραδείγματα. Η εμβάθυνση της ΟΝΕ που είναι υποσυζήτηση αυτή τη στιγμή, απαιτεί αναθεώρηση του ρόλου που παίζουν στατιστικέ στην οικονομική διακυβέρνηση. Η ανάπτυξη των, του, του πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, ο, ε, ο τομέας της ψηφιοποίησης με την ενίσχυση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς ή ο τομέας των μεταναστευτικών πολιτικών απλά παραδείγματα όπου οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα απαιτούν να αναθεωρήσουμε τη, κάποια πράγματα και ούτω ώστε να είναι πιο αξιόπιστες και πιο γρήγορες οι στατιστικές που ετοιμάζουμε. Δεύτερη προτεραιότητα είναι να εστιάσει η Eurostat και να αξιοποιήσει το τρομακτικό ε, δυναμικό που έχουν η ψηφιακή τεχνολογία και οι νέες πηγές. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε πιο γρήγορες στατιστικές, θα έχουμε υψηλότερο επίπεδο λεπτομέρειες για τις περιφέρειες που είναι όλο και πιο σημαντικό, το ξέρετε πολύ καλά αυτό. Ζητάτε και καλά ζητά, κάνετε και ζητάτε κάτι τέτοιο. Ε, να δώσουμε στοιχεία σε επίπεδο όχι απλώς κλασικών ε, περιφερειακών μονάδων, αλλά σε επίπεδο πόλεων ε, για τις παράκτιες περιοχές, για τις διασυνοριακές περιοχές, για περιφέρειες ε, της υπαίθρου κτλ. Και μόνο με τις νέες πηγές και την τεχνολογία μπορούμε να το κάνουμε και να μειώσουμε και το βάρος για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Γιατί οι, επιχειρήσεις, γιατί οι που συλλέγονται θα επαναχρησιμοποιούνται. Τρίτη προτεραιότητα να εστιάσω στον τρόπο με τον οποίο οι επίσημες στατιστικές κοινοποιούνται και διαδίδονται στους χρήστες. Με περηφάνεια σας λέω ότι το τελευταίο χρόνο και όσα ασκούσα τα καθήκοντα της Γενικής Διευθύντριας ε, ξεκινήσαμε ένα, μια εντυπωσιακή οδύσσια να βελτιώσουμε την διάδοση των α, ε, στατιστικών στοιχείων της Eurostat. Είναι η απαρχή του ταξιδιού και τα πρώτα αποτελέσματα είναι προφανή να σας πω τις στάσεις Τι σκοπεύουμε να κάνουμε σε αυτόν τον τομέα. Ξεκινήσαμε τη διαδικασία ανανέωσης της ιστοσελίδας μας, ούτως ώστε να είναι πιο απλή, πιο εύχρηστη και οπτικά πιο ελκυστική. Αρχίσαμε να ετοιμάζουμε ε, ψηφιακές δημοσίευσεις, όχι δηλαδή φακέλους PDF απλώς, αλλά 13 διαδραστικά εργαλεία ε, σε ένα συγκεκριμένο μέρος και ο χρήστης να μπορεί να παίζει με τα στοιχεία, να ξαναχρησιμοποιεί τα στοιχεία, να τα παίρνει, να, παίρνει, να φτιάχνει τις δικές του γραφικές παραστάσεις και αναλύσεις και αυτές οι δημοσιεύσεις επικαιροποιούνται ως αμέσως μόλις συγκεντρώσουμε τα νέα στοιχεία. Ε, ξεκινήσαμε και ένα νέο τμήμα ε, με ειδήσει ε, και θέματα που ενδιαφέρουν τους πολίτες, με ωραία γραφήματα. Ε, και αυτόματα μπορούν να μεταφραστούν σε όλες τις γλώσσες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βελτιώνει την, ε, τη δυνατότητα του πολίτη να καταλάβει αυτά τα νέα. Να σας πω και κάποια νούμερα τώρα, γιατί δεν έχει νόημα να μιλάτε στη Γενική Διευθύντρια χωρίς νούμερα. Πριν από μια εβδομάδα, την Διεθνή ημέρα της γυναίκας, δημοσιεύσαμε με απλό τρόπο ένα γράφημα για την διαφορά ε, μισθών ανδρών και γυναικών μετά αναδημοσιεύτηκε στο Twitter και στο Facebook και για ε, μέσα σε λίγες ώρες τρία εκατομμύρια πολιτών ε, είχαν δει αυτά τα στοιχεία. Πρόεδρε, να σας αναφέρω ακόμα τρία σημεία. Το πρώτο σημείο είναι ότι οι τρεις προτεραιότητες που σας ε, περιέγραψα δεν μπορούν να επιτευχθούν από την Eurostat μόνη. Θα πρέπει να συνεχίσουμε την συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Κοινοβούλιο για να καταλάβουμε τις ε, ανάγκες για πληροφόρηση ακόμα καλύτερα. Η Eurostat δεν παράγει μόνη της τα δεδομένα, τα στοιχεία αυτά. Πρέπει και θα συνεχίσουμε την εταιρική σχέση με τα κράτη-μέλη, ειδικά στο βαθμό που θέλουμε να έχουμε γρηγορότερες στατιστικές, θα ενισχύσουμε τη συνεργασία με, τους το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών και άλλους διεθνείς ε, οργανισμούς. Αυτό είναι το πρώτο, η πρώτη προτεραιότητα. Το δεύτερο σημείο, η δεύτερη προτεραιότητα, θέλω να δράξω την ευκαιρία για να μιλήσω για την ε, επαγγελματική ανεξαρτησία. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να εξασφαλίσω την επαγγελματική ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα των, Ευρω... των Ευρωπαίων στατιστικολόγων και στατιστικών. Εσείς, Πρόεδρε, θεωρήσατε ότι αυτό ήταν προϋπόθεση ε... για την επαγγελματική ανεξαρτησία να μου δώσετε το κατάλληλο νομικό πλαίσιο. Εγώ όμως θα πρέπει κάθε μέρα να παίρνω τέτοιες αποφάσεις ε, για διάφορα θέματα, για τα, τι δημοσιεύουμε στον τύπο, ε, ούτως ώστε οι στατιστικές ε, να είναι αντικειμενικές και γρήγορες. Η επαγγελματική ανεξαρτησία είναι κάτι που θα υπάρχει καθημερινά και θα επιληθώ γι' αυτό. Επανέρχομαι στο θέμα της συνεργασίας. Τους επόμενους μήνες θα έχουμε ποικίλε ευκαιρίε να αποδείξουμε τη θαυμάσια συνεργασία μα. Όπω είπε και ο κ. Γουαλτιέρη, υπάρχουν διάφορες, διάφοροι σημαντικοί νομικοί, νομοθετικοί φάκελοι ε, ή κανονισμοί πλαίσιο που θα διαμορφώσουν τι ευρωπαϊκέ στατιστικέ και που θα πρέπει να υιοθετηθεί συν νομοθετήσει ε, το Κοινοβούλιο για το ΑΕΧ, ε, τη Γεωργία και άλλα θέματα το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Πρόγραμμα για τα επόμενα 7 χρόνια, για το επόμενο ε, πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, θα πρέπει να συμφωνηθεί. Και το Κοινοβούλιο θα παίξει πάλι σημαντικό ρόλο, όχι μόνο για να εντοπιστούν οι ανάγκες για ενημέρωση και πληροφορία, αλλά και να εξασφαλίσουμε ότι οι Ευρωπαίοι στατιστικολόγοι έχουν επαρκείς πόρους στη διάθεσή τους για να κάνουν ακριβώς αυτό που προσδοκούμε. Συμπερασματικά, Βασίζομαι στην συνεχή υποστήριξή σας φυσικά. Παράλληλα όμως χαίρομαι που θα έχουμε αυτό το μόνιμο διάλογο γιατί οι αμοιβαία υποφελείς σχέσεις σημαίνουν ότι προφανώς η Ευρώπη χρειάζεται στατιστικές αλλά η στατιστική μας υπηρεσία χρειάζεται τη συνεχή και απαρασάλευτη υποστήριξή σας. Προσβλέπω σε αυτή τη συνεργασία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ την πολύ αναλυτική σας παρουσίαση. Να. τώρα τον κύριο Κίρτσο από τους συναδελφούς. Ε, very interesting. Πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία. Δύο ερωτήσεις έχω. Η πρώτη σχετίζεται με την σύγκριση των ευρωπαϊκών στατιστικών στοιχείων με τα αμερικανικά. Είναι συγκρίσιμα και τα κινέζικα στατιστικά στοιχεία είναι αξιόπιστα γιατί σε τελική ανάλυση θα τα συγκρίνουμε με τις άλλες μεγάλες οικονομίες. Οπότε τι συμβαίνει σε σχέση με τις ΗΠΑ και την Κίνα. Και μια άλλη συγκεκριμένη ερώτηση, αν σας έχει απασχολήσει το ζήτημα, υπάρχει η λεγόμενη περίπτωση του κυρίου Γεωργίου, ο οποίος ήταν ε, ο διευθυντής ε, της ε, Ελστάτ, κατηγορήθηκε από διάφορους πολιτικούς ότι αύξησε το έλλειμμα έχει απαλλαγεί πολλές φορές στα δικαστήρια αλλά εξακολουθεί να διώκεται κανείς ε, δεν του δίνει πολιτική κάλυψη και ταυτόχρονα ε, η κυβέρνηση έχει συμφωνήσει με τα θεσμικά έργανα ότι το ελληνικό κράτος θα καλύψει τα νομικά του έξοδα. Μια δηλαδή τρελή κατάσταση. Δεν ξέρω αν ε, σας έχει απασχολήσει και αν μπορείτε να μας ενημερώσετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πολύ καλές ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα για την σύγκριση των στατιστικών στοιχείων με τον υπόλοιπο κόσμο, πάρα πολύ σημαντικό. Μια γρήγορη απάντηση είναι ότι η συγκρισιμότητα στατιστικών δεδομένων είναι αποτε, αποτελεί αντικείμενο εγγύησης των ε, κοινών ορισμών, συνήθως υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, όπου η Eurostat και τα κράτη-μέλη συμμετέχουν ενεργά και δεύτερον μέσω άλλων διεθνών οργανισμών όπως το ΔΕΛΤΑ ΩΣΑ και αναλόγως με το θέμα ε, μπορεί να είναι και ο οργανισμός τροφίμων ε, του ΟΗΕ για τα στατιστικά της Γεωργίας. Να σας δώσω ένα πρόσφατο παράδειγμα. Κάθε Μάρτιο έχουμε μία συνάντηση του ΟΗΕ στο Νιούαρκ και η Eurostat, παραδείγματο χάρη, να ανέλαβε μία πρωτοβουλία για στατιστικά στοιχεία για τους πρόσφυγες και ίσως ε, εκπλαγείται, αλλά 70 χρόνια μετά από την σύσταση της Στατιστικής Επιτροπής του ΟΗΕ δεν υπάρχει ένας ορισμός ε, τυποποιημένος του πρόσφυγα. Θέλουμε λοιπόν ε, να, να μπορέσουμε να ηγηθούμε και να έχουμε συγκρίσιμα στατιστικά στοιχεία. Είναι λοιπόν σημαντικό πέρα από τα στοιχεία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουμε συγκρισιμότητα και σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Το δεύτερο ερώτημα αφορά την ε, Ελλάδα. Υπάρχουν κάποια υποερωτήματα. Να πω πρώτα απ' όλα ότι η Eurostat ε, από το 2010 ε, έχει επιβεβαιώσει τα δεδομένα για τα ελληνικά στατιστικά στοιχεία χωρίς καμία επιφύλαξη και αυτό πάντα βεβαίως είναι κάτι το οποίο παραλαμβάνουμε κάθε φορά ότι οι περιπτώσεις όπως οι, αυτές οι οποίες ε, κρεμούν στα δικαστήρια μπορεί να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι δεν είναι έγκυρα τα στατιστικά στοιχεία, κάτι το οποίο δεν ισχύει και το έχουμε πει πολλές φορές. Μετά είχαμε την ε, θέση που έλαβε η αρμόδια επίτροπος και ο αντιπρόεδρος ο κύριος Ντομπρόφσκης και άλλοι επίτροποι. Όσον αφορά τώρα την υπόθεση εις βάρος του πρώην Προέδρου της Ελστατ, βεβαίως ε, παρακολουθούμε την υπόθεση. Και ακολουθώντας βεβαίως τον κανόνα ότι δεν παρεμβαίνουμε στις εθνικές ε, νομοθετικές διαδικασίες, Κάναμε ό,τι μπορούσαμε πέρσι στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την Ελλάδα να τεθούν τα στατιστικά στοιχεία επιτάπητος και οπωσδήποτε καταφέραμε να περάσει ένας νόμος στην Ελλάδα μετά από σύσταση της Κομισιόν για να αποζημιωθεί ο κύριος Γεωργίου για τα δικαστικά έξοδα. Και μπορώ να σας ενημερώσω ότι πράγματι αποζημιώθηκε για τα πρώτα δικαστικά έξοδα. Αυτά είναι τα τελευταία νέα που μπορώ να σας ε, δώσω. Σας ευχαριστώ. Περφάνος Περές. Ευχαριστώ. Καλή τύχη στη θητεία σας εκ μέρους των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Κοινοβούλιο. Ήδη στην εισηγήσή σας δείξατε κάποια σημεία που θα καθορίσουν το διάστημα της θητείας σας. Χθε ήταν εδώ ο πρόεδρος της ΕΣΚΑΔ και επέμεινε πολύ στον τον ανταγωνισμό μεταξύ των στατιστικών ε, φορέων, των κρατικών στατιστικών φορέων και των sexy data provider, των που είναι και και παρέχουν δεδομένα, για να παραφράσω λίγο τα λόγια του. Τέλος πάντων, είναι θέμα που απασχολεί το κοινό, είναι ένα αγαθό κοινό και θα έπρεπε να μπορούν όλα αυτά να διοργανωθούν βάσει των αξιόπιστων στατιστικών που κανονικά διαθέτει η Eurostat. Πέραν όμως της θητείας σας, δεν θεωρείτε ότι πρέπει να υπάρξει κάποια διασύνδεση με την οικονομική διακυβέρνηση της Ευρώπης, λόγω χάρη στο πλαίσιο των συγκεκριμένων αναχώρασεων τάσεων για να είστε βέβαιοι ότι αυτοί από τους οποίους εξαρτάστε, δηλαδή οι Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες, διαθέτουν αρκετά μέσα για να σας τροφοδοτήσουν με τα στοιχεία που χρειάζεστε. Ιδάλλως, ε, κάπου θα πρέπει να τις υποκαταστήσετε και μετά θα αμφισβητηθεί και εσάς η χρηματοδότησή σας, λέγοντας ότι κάνετε τη δουλειά που αναλογεί στους εθνικούς φορείς. Ποια είναι λοιπόν η άποψή σας σχετικά και πώς θα μπορούσαμε να σας ε, βοηθήσουμε κι εμείς για να μην γίνει κάτι το ξεπερασμένο, το βαρετό και το πασέ στατιστική. Αλλά να υπάρχει εξοπιστία σε όλους τους τομείς. Ε, και μια δεύτερη ερώτηση, επειδή εντοπίσατε κάποια σημεία όπου είναι καθοριστική σημασία να έχουμε αξιόπιστα στατιστικά δεδομένα, αλλά το κοινωνικό είναι μείζον θέμα. θέλετε την κοινωνικό πυλώνα και εδώ ενθυμούμε ότι όταν μιλάμε για θέματα απασχόλησης δημιουργείται ένα παράδοξο, διότι τα διευθυντικά ταμεία προβλέπονται και δεσμεύονται ανάλογα με τις περιοχές που ονομάζονται needs τρία Ε, και, ε, και η απασχόληση καταμετράται ένα περιοχή. Πώς όμως γίνεται αυτό αναχώρα βάσει των περιοχών ΝΑΤΣ 3 και μετά θα μπορούσατε να μας δώσετε στατιστικά δεδομένα ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιδιώξει τους στόχους της της COP21 και της σχετικής συμφωνίας. Ευχαριστώ κύριε Μπερές. Θα συνεχίσω αγγλικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Ε, γνωρίζω ότι βεβαίως ε, θα χρειαστώ στήριξη στους δύσκολους αυτούς ε, καιρούς. Η παρέμβασή σας κάλυψε αρκετά σημαντικά ζητήματα. Θα προσπαθήσω να εστιάσω στην απάντησή μου γιατί θα συνεχιστεί ο διάλογος μας. Ναι, πρέπει να δούμε το θέμα των ανταγωνιστικών παρόχων υπηρεσιών. Τώρα, αν κάτι τέτοιο είναι άδικο, είναι μια καλή ερώτηση, αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε και να παρακολουθούμε το τι συμβαίνει. Και μια σημαντική πτωχή, πτυχή την οποία τονίζω ε, μιλάμε για το ανταγωνιστικό κομμάτι, πρέπει να είμαστε και πιο γρήγοροι και πιο αξιόπιστοι. Όσον αφορά το θέμα της εμπιστοσύνης, πρέπει να το κερδίσουμε. Δεν σημαίνει ότι είναι δεδομένο ότι ο κόσμος θα προτιμάει τη Eurostat και τα επίσημα στατιστικά στοιχεία. Όσον αφορά δε τις συστάσεις αναχώρα, το τι μπορείτε να κάνετε για να μας βοηθήσετε θα έλεγα να είστε ο εαυτό σας. Ε, συνεχίσετε να λέτε ότι τα ευρωπαϊκά στατιστικά στοιχεία πρέπει να είναι στην συζήτηση ευθύς εξ αρχής όταν μιλάμε για εμβάθυνση της ΟΝΕ για την διανομή των κονδυλίων που τα επόμενα χρόνια θα έχουν μία αιρεσιμότητα και το θέμα είναι ακριβώς πώς να μετρηθεί αυτή η αιρεσιμότητα και εκεί πέρα γύρεται το θέμα των στατιστικών στοιχείων. Οπότε υψώστε την φωνή σας ότι πρέπει να είμαστε εκεί ευθύ εξ αρχής για το πώς θα μετρηθούν αυτά τα φαινόμενα. Μετά υπάρχει ένας τρόπος ε, για να λάβετε κι εσείς μέρος. Έχετε τώρα κάποιους κανονισμούς επιτάπητος ε, και ε, έχουμε την εντύπωση ότι μας στηρίζεται στον τριμερή διάλογο μεταξύ ε, Κομισιών, Κοινοβουλίου και Κρατών Μελών, γιατί τα χρειαζόμαστε τα κράτη-μέλη ε, και δεν είναι μόνο θέμα πόρων, αλλά πρέπει ακριβώς να κινηθούμε γρηγορότερα και πρέπει να δούμε ακριβώς αυτή την πλατφόρμα. Εντάξει, γενικά είναι συντηρητικοί οι στατιστικολόγοι, αλλά πρέπει να κινηθούμε γρήγορότερα, να χρησιμοποιήσουμε νέες πηγές ε, όταν ε, συζητάμε και τον ε, κανονικό πλαίσιο. Βεβαίως, ιστορικά τα στατιστικά στοιχεία για την οικονομία ήταν τα σημαντικότερα. Τώρα υπάρχουν βεβαίως και τα περιβαλλοντικά και τα κοινωνικά. Πρώτα απ' όλα είναι το θέμα του χρονισμού. Ξεκινήσαμε πέρυσι και ακούτε πάρα πολλά πράγματα ε, και για τα κοινωνικά, τις ε, συνθήκες ε, ζωής, αλλά κάτι μπορεί να γίνει. Επίσης αναφέρατε το θέμα του περιφερειακού επίπεδου και βεβαίως ε, τρόπος για να ε, προχωρήσουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε και εδαφικές ε, πληροφορίες για μεγαλύτερο επίπεδο ανάλυσης. Και για το μέλλον, για την COP 2020, και αυτό είναι στην ημερήσια διάταξη, όπου έχουμε έναν αριθμό νέων δικτών για τη συλλογή προφοριών. Οπότε η συμβουλή μου αυτό θα ήταν, να είστε ο εαυτός σας. Και να τονίζετε ότι χρειάζονται τα δεδομένα. Σας ευχαριστώ. Το ECR τώρα. Σας ευχαριστώ, κυρία Διευθύντρια. Όταν μιλάμε για τα ευρωπαϊκά στατιστικά στοιχεία, η ομάδα μας θεωρεί ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να τηρήσουμε την αρχή της επικουρικότητας. Και βεβαίως ε, έχουμε και τον κανονισμό του 2012, ο οποίος είχε προσπαθήσει να ενισχύσει την ανεξαρτησία αυτήν ενισχύοντας ε, την αυτονομία των εθνικών υπηρεσιών. Μπορείτε να αξιολογήσετε τον αντίκτυπο αυτών των αλλαγών στην δουλειά της Eurostat. Εσείς θεωρείτε ότι η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών υπηρεσιών και της Eurostat έχει βελτιωθεί είναι πιο συγκεκριμένα, πιο αξιόπιστα ή είναι χειρότερη τώρα η κατάσταση. Βλέπετε κάποια διαφορά. Και θεωρείτε τώρα ότι οι εθνικές υπηρεσίες εμπλέκονται περισσότερο στο πώς λειτουργεί η όλη η διαδικασία. Και πώς μπορεί να βελτιωθεί η ολη διαδικασια και πως μπορει να βελτιωθει η νομοθεσια σας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την σημαντική πτυχή των σχέσεων της Eurostat με τα κράτη-μέλη. Ο κανονισμός ε, για τα στατιστικά στοιχεία άλλαξε για να ενισχυθεί πραγματι η επαγγελματική ανεξαρτησία και βεβαίως είχαμε ακριβώς το θέμα της ενίσχυσης της εμπιστοσύνης ε, και των συστάσεων που γίνονται από την εξέταση από συναδέλφους και ομοτήμους και ακριβώς αυτά θα φανούν όσον αφορά και την εφαρμογή των συστάσεων αυτών των διαδικασιών και την υποβολή της σχετικής έκθεσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις αρχές Ιουνίου. Όσον αφορά την εφαρμογή του νόμου, βεβαίως θα την παρακολουθούμε και είμαι πεπισμένη ότι αυτή είναι η κοινή αντίληψη των ε, διευθυντών ε, των εθνικών ε, υπηρεσιών, ότι αυτές οι αλλαγές στην νομοθεσία έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της θέσης των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών, γι' αυτό ακριβώς υπάρχει ο δικός σας ο ρόλος. όσον αφορά την σχέση με τα κρατημέλη, με τιμή η εμπιστοσύνη των Προέδρων των Εθνικών Στατιστικών Υπηρεσιών και έχουμε μια εντατική συνεργασία γιατί αντιμετωπίζουμε και κοινέ προκλήσεις. Όχι μόνο η Eurostat, όλες οι στατιστικές υπηρεσίες έχουν τις προκλήσεις των νέων τεχνολογιών, των ανταγωνιστών, μείωση να, να, η πίεση να μειωθεί το βάρος, να χρησιμοποιήσουμε νέες πηγές και να βρούμε κάποιες κοινέ προτεραιότητες για τα επόμενα 7 χρόνια. Οπότε νομίζω ότι θα έχουμε μια καλή συνεργασία με τα κράτη-μέλη και έτσι θα προχωρήσει το θέμα των ευρωπαϊκών στατιστικών στοιχείων γιατί όπως είπαμε αυτά παραγόνται σε εθνικό επίπεδο σε συνεργασία με τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες. Σας ευχαριστώ κυρία Αγγύρνικ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τρει ερωτήσει. Πρώτον, πιστεύετε ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωση για την ακρίβεια και την έκδοση των δεδομένων για το χρέο και το έλλειμμα των κρατών μελών στα πλαίσια του Συμφώνου Σταθερότητα και Ανάπτυξη. Δεύτερον, Υπάρχει ενδεχομένως έλλειψη από εμπιστοσύνη ε, μεταξύ των κρατών μελών, των στατιστικών του υπηρεσιών και τη Eurostat επηρεάζει αυτό την πρόσβασή σα στι πληροφορίε που είναι απαραίτητε για την εκτέλεση των καθηκόντων σα. Και τέλο, με την παράταση του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Προγράμματο, το Κοινοβούλιο ε, Θεώρησε ότι πρέπει να συμπεριληφθούν και άλλοι τομεί και όχι μόνο αυτοί που ορίζονται στι 10 προτεραιότητε ε, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο κείμενο GDP and Beyond. Ποια είναι η άποψή σα για αυτή τη δυνατότητα να προχωρήσουμε για να αυξηθεί το σύνολο των στατιστικών δεδομένων και των μελετών που μπορεί να προκύψουν. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ κυρία Βίρνη για, την, ε, για τις πολύ συγκεκριμένε και εξειδικευμένε ερωτήσεις σας. Πρώτα απ' όλα να πω ότι το χρέος και οι στατιστικές για τα ελλείμματα είναι ο τομέας όπου οι στατιστικολόγοι επενδύουν τα μάλα για να είναι βέβαιο ότι υπάρχει ακρίβεια. Είναι ο μόνος τομέας όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σχεδόν ε, δυνατότητες ε, λογιστικού ελέγχου όπως προβλέπει ο νόμος. Στα κράτη-μέλη και πηγαίνουμε και κοιτάζουμε τους λογαριασμούς και τα βιβλία τους και επαληθεύουμε το πόσο μεγάλες δαπάνες των κυβερνήσεων και των κρατικών φορέων κατηγοριοποιούνται και ούτω καθεξής. Ούτω καθεξής. Είναι ένα καθήκον αρκετά βαρύ. Ε, κάθε φορά που εκδίδουμε τέτοιε στατιστικές, εξασκούμε από τις αρμοδιότητες μας με πλήρη επαγγελματισμό, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι υπάρχει σταθερότητα. Βεβαίω, η ακρίβεια ίσως να μην είναι το πρώτο που μας απασχολεί το κατά πόσο είναι εύστοχα τα δεδομένα μας, μας απασχολεί κυρίω, δηλαδή στην οικονομική διακυβέρνηση και την εμβάθυνση της Νομισματικής Ένωσης. Καθώς συζητάτε τώρα και το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, το πρόβλημα είναι το πεδίο, το θέμα είναι η συχνότητα και το περιεχόμενο. Εάν οι στατιστικές, τα στατιστικά δεδομένα που συλλογούμε είναι κατάλληλα για τον σκοπό τους. Δηλαδή, το ερώτημα είναι αν αυτά που συλλέγουμε είναι εύστοχα, αν ε, συλλέγονται γρήγορα και αν ε, εξυπηρετούν το σκοπό των μελλοντικών μεταρρυθμίσεων. Ω προ του κρατικού φορεί των καταμελών, ε, η απάντησή μου είναι όχι. Δεν αισθάνομαι καμία απειλή, κανένα κίνδυνο, καμία επιφυλακτικότητα από πλευρά των κρατομελών. Αυτό εν μέρη το απήντησα και στο προηγούμενο σύνολο ερωτήσεων. Έχω την αυτοπεποίθηση ότι έχουμε καλή εταιρική σχέση Ας πούμε, πώς, ε, το ερώτημα είναι πώς μοιράζουμε τους συνεργάτες μας μεταξύ γύρω στα 100 μελών για να έχουμε την καλύτερη δυνατή απόδοση. Ως προς το τα όσα υπόθηκαν στο GDP and beyond ε, και επειδή υπήρξα υπεύθυνη Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας και διεύθυνα πολύ κόσμο, να πω ότι πολλά έχουν γίνει και από τη γύρω και από τα κάτι μέλη για να συμπληρώσουμε το, τα στοιχεία του ΑΕΠ με δείκτες συγκριτική αξιολόγηση για την ποιότητα ζωή, για το περιβάλλον, με δείκτες για την κατανομή του εισοδήματο. Τώρα τις πληροφορίες αυτές θα συνεχίσουμε να τις ε, συλλέγουμε και να τις μελετούμε, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τους στόχους του 2030 ή ε, αυτούς της βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτέ οι εξέλιξει πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, όπω και η κεκλική οικονομία ή η COP21 ή το βαθμολόγιο και οι υποκείμενοι δείκτε που θα είναι σημαντικοί για τη λήψη αποφάσεων σε αυτού του τομεί. Συνεχίζουμε πάντως την ίδια πορεία, ακολουθούμε την ορμή που μα έχει δώσει το GDP and Beyond και συλλέγουμε στατιστικά δεδομένα για να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκε των πολιτικών πρωτοβουλειών. Πρόεδρος, ευχαριστούμε ο κύριος Γκίγκολτ. Ευχαριστώ. Κατά πρώτον και από εμά συγχαρητήρια για τον διορισμό σας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Γιατί πάντα πιστεύαμε ότι είσαστε άνθρωπος των πράξεων και αυτό που μας άρεσε. Το εκτιμούμε αυτό. Ε, έχουμε σοβαρές ανησυχίες για αυτή την ιστορία στην Ελλάδα. Δεν έχει ξανασυμβεί ένας στατιστικολόγος να συλληφθεί ε, γιατί το αποφάσισαν ε, οι δικαστικές αρχές και επειδή υπήρχε αμέλεια από τους πολιτικούς. Θέλουμε να προσκαλέσουμε για δεύτερη φορά τον κύριο Γεωργίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ούτω ώστε να κρατήσουμε την πίεση στην Ελλάδα. Η αόριστη απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην γραπτή μας ερώτηση για αυτό το θέμα είναι ντροπή. Δεν ξέρω αν η Κομισιόν εκπροσωπείται, αλλά όταν συμβαίνει αυτοί που ενημερώνουν το κοινό για τα αποτελέσματα ε, να συλλαμβάνονται και να αντιμετωπίζουν ε, τέτοιους κινδύνους, δεν μπορούμε να έχουμε στατιστικό σύστημα. Ε, ξεπεράστηκε μία κόκκινη γραμμή εδώ. Για τη μελλοντική μας σχέση θα ήθελα να κάνω μία πρόταση και εσείς μπορείτε να το λάβετε υπόψη σας. Όπως ξέρετε, Έχουμε το στατιστικό μας πρόγραμμα και υπήρξε κάποια συνέχεια, κάποια δυσαρέσκεια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο παρελθόν, κάποια στοιχεία του στατιστικού προγράμματος δεν υλοποιήθηκαν. Ξέρετε την ιστορία αυτή και ίσως χρήσιμο θα ήταν να έχουμε ένα état de ε, ένα κατάλογο δηλαδή ε, με τα στοιχεία ε, όπου θα βλέπουμε πόσο μακριά έχετε πάει πριν από την ε, τακτική μας συνάντηση για τα κοινωνικά θέματα, για τα περιβαλλοντικά θέματα και, τη, και την παραγωγή στατιστικών. Εσείς για αυτά τα θέματα μας υποστηρίξατε στις διαπραγματεύσεις, αλλά καλό θα ήταν να υπάρχει μια ετήσια έκθεση και μετά από την ανταλλαγή απόψεων να ετοιμάσετε μια σύντομη έκθεση για να μας πείτε ποια από τα νέα στοιχεία του προγράμματος έχουν προχωρήσει, πού έχουν φτάσει, τι προβλήματα αντιμετωπίσετε και να μας βοηθήσετε και εμάς ως νομοθέτες και διατάκτες του προϋπολογισμού να σας δώσουμε τα μέσα. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξη και για το ενδιαφέρον Με αυτή την υποστήριξη συνειδητοποιούμε ότι έχουμε σημασία και καταλαβαίνουμε και πού πρέπει να βελτιωθούμε. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε διάλογο που να βασίζεται σε συγκεκριμένα πράγματα. Γι' αυτό ακριβώ κάνουμε και αυτή τη συζήτηση. Πολύ ωραία. Για το διάλογο σας, σας ρώτησα, μήπως θα μπορούσαμε να έχουμε αυτό το θα μπορούσαμε να έχουμε αυτό το συγκεκριμένο κείμενο. Ε, θα το συζητήσω με τον κύριο Γκουαλτιέρη για να δω ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να συνοψίσω αυτό το, να ετοιμάσω αυτό το, το σύντομο κείμενο, ας πούμε. Θα μπορούσαμε να το βάλουμε ε, ως σημείο προς συζήτηση στους συντονιστές για να δούμε τι εναλλακτικέ υπάρχουν, να το συζητήσουμε και να αποφασίσουμε. Καλημέρα, θα μιλήσω πορτογαλικά Θα ήθελα να θέσω δύο ερωτήσεις. Η μία είναι γενική και η άλλη πιο συγκεκριμένη. Η γενική είναι να μας πείτε κάτι παραπάνω για την διακυβέρνηση, το πώς ε, διαχειρίζεστε τη Eurostat. Δηλαδή, κατάλαβα ότι είναι ζωτική σημασίας να ε, συνδυάσουμε τη ζήτηση πληροφοριών από τα θεσμικά όργανα, από τους πολίτες, από τους δημοσιογράφους, να τη συνδυάσουμε με την προσφορά πληροφορίας, που στην ουσία είναι αυτό που παράγει η Eurostat. Για να βρούμε το σημείο ισορροπίας ε, σε αυτήν την προσπάθεια πώς ε, συνδυάζονται οι δραστηριότητε της Εκτελεστικής Επιτροπής ή των Εθνικών Στατιστικών Συστημάτων. Πώς γίνεται η αποτίμηση αυτής της διαδικασίας. Πώς βλέπουμε αν μπορεί να βελτιωθεί όταν προκύπτει κάποια ανάγκη σε επίπεδο κοινωνικού πυλώνα ή οποιαδήποτε άλλη. Πώς η, όλη, ο όλος μηχανισμός της στα προσαρμόζεται πώς γίνεται η διαβούλευση και πώς λαμβάνονται αποφάσεις για να αποδοθούν τα κονδύλια στις ε, ανάγκες που εντοπίζουν. Αυτή ήταν η πρώτη ερώτηση. Η δεύτερη, που είναι πιο εξειδικευμένη και έχει σχέση με την προηγούμενη βεβαίω, είναι ότι είναι, πολύ, είναι θέμα συγκεκριμένων μαθηματικών υπολογισμών βέβαια, αλλά είναι ένα πρόβλημα που έχει απασχολήσει πολύ το Κοινοβούλιο. Φορολογική απάτη. Υπήρξε και ειδική επιτροπή, εξεταστική επιτροπή που εξέτασε το θέμα αυτό εντελεχώ και μας εγείρει δύο προβληματισμούς. Πρώτα απ' όλα την ανάγκη περισσότερων πληροφοριών για να μπορέσουμε να διερευνήσουμε καλύτερα αυτό το φαινόμενο και το άλλο, η άλλη πτυχή που προκύπτει με όλη αυτή τη δουλειά έχει καταλήξει στην παραγωγή περισσότερων πληροφοριών λόγω χάρη ε, με διάφορα έγγραφα των ε, πολυεθνικών εταιριών είδαμε ότι εξαιτίας των, ανα, των ειδικών αναχώραση στάσεων και όσων προέκυψαν με την ε, διερεύνηση της προαπάτης για τις πολυεθνικές είναι πολύ περισσότερα τα έγγραφα που δημοσιοποιούνται. Μιλάμε για πληροφορίες που τώρα ε, προκύπτουν και είναι και καρπός και παράγωγο της νομοθεσίας που συζητάμε και σχεδιάζουμε. Thank you very much, Mr. Ευχαριστώ κύριε Βιέγας. Μίλησατε για τόσα πολλά θέματα. Βλέπετε πόσο ενδιαφέρουσα είναι αυτή η δουλειά. Μετά από ένα χρόνο από την τελευταία συνέντευξη με ρώτησαν ε, αν εξακολουθώ να θέλω τη δουλειά αυτή μετά από ένα χρόνο εμπειρίας. Ένα λόγο που είπα ναι είναι ότι πραγματικά με ενδιέφερε. Είναι εντυπωσιακή δουλειά γιατί μπορεί να δώσει κάτι απτό μετά από, αφού αντιμετωπίσει πολλές προκλήσει και πολλές δυσκολίες. Λοιπόν, ας προσπαθήσω να σα απαντήσω στα πολύ άριθμα σημεία που αναφέρατε. Όντω, μίλησατε για ένα πολύ κεντρικό θέμα. Ε, η ζήτηση και προσφορά. Για τη ζήτηση. Έχουμε μία διαδικασία συλλογής των ετοιμάτων διαφόρων χρηστών. Ε, Παραδείγματο χάρη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, των διαφόρων υπηρεσιών τη της ε, Κομισιόν. Από εκεί ξεκινάμε, έτσι, από αυτού τους χρήστες. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Στατιστική Συμβουλευτική Υπηρεσία, που είναι εκπρόσωποι των ε, ε, οργανώσεων των επιχειρήσεων, ε, των ΜΜΕ, των ερευνητών ε, του Κοινοβουλίου, διαφόρων ομάδων χρηστών δηλαδή. Οπότε κάνουν μια διαβούλευση μαζί τους και εν συνεχεία Έχουμε μια δημόσια διαβούλευση, όπω λέει και η Κομισιόν, όπου οι πολίτες επίσης μπορούν να θέσουν κάποια θέματα Κοιτάμε όλα αυτά τα αιτήματα και μετά ξεκινάμε τη συζήτηση με τα κράτη-μέλη. Γιατί η Eurostat από μόνη τη δεν ετοιμάζει τα νούμερα. Τα νούμερα τα, μα τα δίνουν τα κράτη-μέλη. Και με ρωτάτε πώς μπορώ να αξιολογήσω την κατάσταση. Ε, το θέμα είναι όλο και πιο πολύ θέμα πόρων. Είναι θέμα επιλογών. Πρέπει να θέσουμε προτεραιότητε. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό σε αυτή τη συζήτηση τα εθνικά οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες να μην είναι μόνες τους, να γίνει και μια συζήτηση εθνικά. Ε, όλα αυτά που εμείς απαιτούμε ως Κοινοβούλιο, ως ε, Eurostat, να μας, να τα υποστηρίζει, να υποστηρίζει δηλαδή και, το εθνικό επίπεδο. Δεύτερον, εσωτερικό, ένα, υπάρχει ένα εσωτερικό επίπεδο. Ε, κάνουμε έναν επικοδομητικό διάλογο αλλά θα πρέπει να βρίσκουμε όλο και περισσότερο λύσει. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με τι έρευνε όπω κάναμε παλιά, γιατί είναι πολύ ακριβέ, είναι ε, πολύ επαχθεί και πρέπει να χρησιμοποιούμε άλλους, άλλες πηγές, ας πούμε διοικητικές πηγές. Γι' αυτό ε, το βασικό ερώτημα για την παραγωγή στοιχείων είναι πώς θα χρησιμοποιήσουμε νέες πηγές. αυτό είναι βασικό ερώτημα ε, το πώς θα θέσουμε δηλαδή τις προτεραιότητες. Είναι ερώτημα κλειδί, ούτως ώστε να είμαστε αποτελεσματικοί. Θα πρέπει να έχουμε και τους κατάλληλου πόρους, αλλά θα πρέπει να έχουμε και ένα σύστημα που θα μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε απο, ε, αποτελεσματικά τους, ε, τις πηγές. έπειτα, ε, με τον κύριο Γκίγκολτ και τον κύριο Γκουατιέ συζητήσαμε το θέμα της φοροδιαφυγής και ξέρω ότι είναι σημαντικό για το Κοινοβούλιο. Το θέμα είναι τι είναι ευθύνη το, της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας. Δεν είναι δική μας αρμοδιότητα να, να αποφασίσουμε και να αντιμετωπίσουμε τη φοροδιαφυγή, αλλά το να μετρήσουμε την οικονομία, διάφορα οικονομικά μεγέθη. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, ας πούμε, η ψηφιοποίηση και η επιμερισμένη οικονομία. Τίθεται το θέμα του ρόλου των ε, ενδιαμέσων εταιριών όπως, ας μην πω ονόματα τέλος πάντων, που προσφέρουν υπηρεσίες ε, ίντερνετ. Το βασικό ερώτημα είναι αν θα πρέπει οι δραστηριότητε του να φορολογούνται ή όχι. Αυτό είναι δική σα δουλειά. Εσεί θα το αποφασίσετε. Εμεί θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι έχετε τι πληροφορίε για το μέγεθο και το τι παράγεται. Πόσα άτομα εργάζονται εκεί, έτσι τα λέω απλοϊκά τώρα. Θα πρέπει να σας δώσουμε πληροφορίες που σας επιτρέπουν να παίρνετε αποφάσεις για τα θέματα της φοροδιαφυγής. Τέλος, αναφέρατε τις εκθέσεις των επιμέρους κρατών μελών. Αυτό πρέπει να το ε, τονίσω ότι υπάρχει μια αλλαγή εδώ σε σχέση με το παρελθόν. Ε, στο παρελθόν αναφερόμαστε σε, σε, στα σύνολα, σε σωρευμένα νούμερα. Ε, τώρα θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένες συγκριτικές στατιστικές χωρών. Είναι και θέμα επιμερισμού εργασία. Να έχουμε μια συνεργασία με τι εθνικέ στατιστικέ αρχέ αφενός, να διαδίδονται οι στατιστικέ, ε, δηλαδή να μα στέλνουν τι στατιστικέ τους και πρέπει να μα βοηθήσουν για να διαδίδουμε τα στατιστικά στοιχεία που παράγουμε τα παράγουμε εμεί, αλλά πρέπει να διαδίδονται με συνεχεία σε εθνικό επίπεδο. Γιατί θα πρέπει να ε, περιγράφονται και αυτά τα νούμερα και στη γλώσσα, τη της κάθε χώρας πια. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σίλβα Περέιρα. Ευχαριστώ. Και εγώ πορτογαλικά θα μιλήσω. να καλωσορίσω τη Γενική Διευθυντρία της Eurostat και να επιβεβαιώσω ότι, όπως είπατε, η σημασία των ε, καλών στατιστικών που θα μας φτάνουν εγκαίρως και θα μπορούν να είναι συγκρίσιμες ε, είναι σημαντική για να μπορεί η κοινωνία να κατανοήσει την οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα και για να ληφθούν αποφάσεις τεκμηριωμένες ε, όχι μόνο από, τους δημόσ, από τις δημόσιες αρχές αλλά και από τους οικονομικούς παράγοντες και μετά να μπορεί κανείς ε, με τα λόγω γνώσεως να λάβει τις σχετικές του αποφάσεις. Θέλω λοιπόν να θέσω δύο ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα η ταξινόμηση των ε, μέτρων που είναι έκτακτα, τα one-off, που είναι μια στατιστική ε, δραστηριότητα πολύ σημαντική για την οικονομική διακυβέρνηση. Νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου. Έχουμε εδώ δύο προβλήματα. Πρώτα απ' όλα είναι η καθυστέρηση στην ταξινόμηση αυτών των στατιστικών δραστηριοτήτων. Υπάρχουν περιπτώσεις που εδώ και μήνες σέρνονται, κάποιες φορές ακόμη και παραπάνω, για να δούμε αν τελικά ένα μέτρο πρέπει να ταξινομηθεί ως έκτακτο ή όχι. Στην Πορτογαλία, λόγου χάρη, εδώ και μήνες γίνεται κουβέντα μεταξύ της Eurostat, της στατιστικής μας υπηρεσίας και του Υπουργείου Οικονομικών για το κατά πόσο θα κεφαλαιοποιηθεί η Kaiser General Depositus, η Γενική Τράπεζα Καταθέσεων. Ε, και σε τι κατηγορία θα μπει το μέτρο αυτό. Η καθυστέρηση αυτή προφανώς δημιουργεί προβλήματα. Το ερώτημα λοιπόν είναι τι μπορεί να γίνει για να συντομεθεί αυτό το διάστημα εντός του οποίου μπορεί να ληφθεί μια απόφαση. Και επίσης τι υποκρύπτει αυτή η καθυστέρηση. Μήπως υποκρύπτει κάτι το ε, σκοτεινό ή αδιαφανές ως προς τους κανόνες Δηλαδή δεν βγάζει νόημα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι στατιστικές υπηρεσίες, οι κυβερνήσεις, όλοι να ερμηνεύουν διαφορετικά τους κανόνες και οι κυβερνήσεις να πρέπει να λάβουν πρώτα αποφάσεις και μετά να περιμένουν να βρεθούν σε στάση αναμονής για να δουν τι θα πούν οι στατιστικές υπηρεσίες. Αυτό θα πει ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα σαφήνειας των κανόνων ε, ως προς την ταξινόμηση μιας έκτακτης δραστηριότητας. Ε, ή την ταξινόμηση της ως έκτακτης ή όχι. Εδώ λοιπόν με ενδιαφέρει τι μπορεί να κάνει η Eurostat ώστε να λαμβάνονται αποφάσεις αφέστερες με κανόνες πιο εύληπτους ώστε να μπορούν όλοι και τα της οικονομικής διακυβέρνησης να ε, οργανωθούν βάσει αρχών που να είναι κατανοητές με τον ίδιο τρόπο σε όλους. Ευχαριστώ κύριε Περέιρα. Αυτό το σύνολο ερωτήσεων είναι πολύ σημαντικές και είναι μια ευκαιρία να απαντήσω σε κάτι που δεν έχει άμεσα σχέση με το έργο της στατιστικής αυθυρός. Αυτό που είπατε έχει να κάνει με το πώς στατιστικώς κάποιες δραστηριότητες μπορούν να ταξινομηθούν. Να πω κατά πρώτον ότι συμφωνώ απολύτω. Οι κανόνε πρέπει να είναι σαφεί και εύληπτοι. Πρέπει να υπάρχει προβλεψιμότητα και πρέπει να είναι και διαφανεί. Ε, γι' αυτό Πέρυσι, όταν ορίστηκα, ασκούσα τα καθήκοντα Γενικού Διευθυντή αρχικά, μια από τις πρώτες μου ένα από τα πρώτα μου μελήματα ήταν να προβλέψω κανόνες για τέτοιες περιπτώσεις. Κανόνες για το τι θα ισχύει σε αυτές τις περιπτώσεις, σε τι χρονικό όριο θα γίνονται όλα, πότε θα συζητιόνται και πότε θα υλοποιούνται σχετικέ αποφάσει. Διότι πρέπει να υπάρχει κάποια διαφάνεια και αρκετό χρόνο ώστε οι στατιστικέ υπηρεσίε να μπορούν να εφαρμόσουν του κανόνε. Έπειτα, κάτι που θεωρώ σημαντικό και ξεκινήσαμε να το κάνουμε πέρσι και αυτή την κατεύθυνση ακολουθούμε ακόμα, είναι ότι επί σειρά ετών υπήρχε η ιδέα ότι η στατιστική αντικατοπτρίζει και καταγράφει μόνο ότι έχει συμβεί. Τώρα θέλουμε να δώσουμε έμφαση στο σκέλος της πρόληψης, ιδίως για μεγάλα επενδυτικά προγράμματα ή έργα και για μεγάλες στατιστικές δραστηριότητες εφόσον τις αναμένουμε. Γιατί λαμβάνει όλο ένα και μεγαλύτερη σημασία για τους επενδυτές λόγω χάρη στα πλαίσια του ΕΦΣΥ, του επενδυτικού προγράμματος για την Ευρώπη, να γνωρίζουν όχι μόνο τους κινδύνου και τα ωφέλη, αλλά επίσης να γνωρίζουν πώς θα χαρακτηριστούν στατιστικώς οι διάφορες ε, δράσει και ενέργειες Γι' αυτό σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, ε, έχουμε σχεδιάσει και σε συνεργασία και με τους υπευθύνους των κρατών μελών, με όσους σχεδιάζουν χρηματοοικονομικά εργαλεία και με τραπεζικού κοιτάζουμε να δημιουργήσουμε ένα σύνολο μεθοδολογικών εργαλείων για τα βασικά χρηματοπιστωτικά εργαλεία, όπω τι ε, εταιρικέ σχέσει δημόσιο ιδιωτικού τομέα, όπω τι ενεργειακέ συμβάσει ή τι παραχωρήσει. Εδώ κοιτάζουμε πώς στατιστικώς αυτά τα νέα χρηματοπιστωτικά εργαλεία θα μπορούν να ταξινομηθούν σωστά. Και αρχίσαμε τις μεθοδολογικές αυτές συμβουλές να τις αποστέλνουμε σε όλους τους ενδιαφερομένους. Δηλαδή μπορεί κανείς να έρθει από πριν να περιγράψει την οικονομική δραστηριότητα που προβλέπει να κάνει ε, Συνήθω πάνε στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, αλλά αυτά μπορούν να απευθούν και στη Eurostat και μετά του λέμε αν συνάδουν με του κανόνε μα. Ε, φροντίζουμε να έχουμε συνομιλίε με ομάδα περιεχομένων από τα κράτη-μέλη, ώστε να υπάρχει ισότιμη μεταχείριση όλων στι ίδιε οικονομικέ δραστηριότητε και ε, προσφέρουμε συμβουλευτική ουσιαστικά για να υπάρχει η σωστή καθοδήγηση και να είμαστε και διαφανείς. Και όλες οι αποφάσεις για τη στατιστική μεταχείριση βάσει αιτήματος ε, κράτους μέλους, δηλαδή ως ε, εκ των προτέρων συμβουλή, να μπορεί να προσφερθεί και επίση να δημοσιευθεί και στον ιστότοπο της Eurostat ώστε να είναι διαφανή τα πάντα και όλοι να μπορούν να ωφεληθούν από αυτό. Εδώ θίξατε δύο σημεία αρκετά ε, λεπτά τα οποία θέλω να τα ε, σχολιάσω. Γνωρίζω την περίπτωση τη Πορτογαλία γιατί ξέρω πολύ καλά τι συμβαίνει στη Γύρω Στάτ και αναφέρεστε σε αποφάσει που συνήθω, θα Δεν είναι η ίδια η μεταχείριση της Γενικής Διεύθυνσης ε, Ανταγωνισμού, θεωρώντας αν κάποια ε, δραστηριότητα είναι κρατική βοήθεια ή όχι και δεν είναι η ίδια αξιολόγηση της Eurostat που χρησιμοποιεί άλλα κριτήρια. Δεν είναι δική μας λοιπόν δουλειά να χαρακτηρίσουμε αυτό το μέτρο, αλλά είναι περισσότερο οι συνάδελφοι του ΕΚΦΙΝ που πρέπει να ταξινομήσουν αυτή την ε, συναλλαγή, αυτή την, εμπορική, την οικονομική ε, δραστηριότητα. Πρέπει να δούμε κυρίως εμείς τι ε, ποσό ελλείμματος υπάρχει και αν ε, είναι συγκεκριμένο και ακριβές το ποσό. Πάντως, ναι, έχουμε ενισχυμένο ρόλο να προλαμβάνουμε τέτοιες περιπτώσεις, να προσφέρουμε συμβουλές, να είμαστε διαφανείς, να είμαστε ταχύτεροι για τα νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία και αυτό στα πλαίσια γενικότερα της οικονομικής διακυβέρνησης. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Σόρου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη που έχω αυτή τη βραχνή φωνή. Κυρία Διευθύντρια, μα μιλήσατε για τι μεγάλε τεχνολογικέ αλλαγέ που επηρεάζουν την δραστηριότητα και τον τρόπο που παράγονται οι στατιστικές. Ε, θα θυμάστε πώς γίνονταν στο παρελθόν. Τώρα έχουμε το, την εκμάθηση μηχανής ε, και όλα αυτά τα πράγματα, τα ψηφιακά. Υπάρχουν και άλλες σημαντικές κοινοτομίες, αν όχι πιο σημαντικές, για τη συλλογή των δεδομένων σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους που ήταν οι δημοσκοπήσεις, οι ε, η έρευνα, ε, που κάναμε μέσω επιχειρήσεων και σε ιδιώτες. Τώρα έχουμε τις μεγάλες πλατφόρμες του ίντερνετ που μας δίνουν ατέλειωτα δεδομένα, άπειρα δεδομένα. Που, που συνήθως ε, δεν συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των πηγών ε, της ε, Eurostat και των Εθνικών Στατιστικών Υπηρεσιών. Για αυτό το θέμα... Το Κοινοβούλιο έχει μιλήσει. Υπάρχει και μια έκθεση πρωτοβουλίας για την οικονομία που βασίζεται στα δεδομένα. Ε, κάναμε και μια έκθεση επίσης για την καινοτομία και τα όρια της τεχνολογικής, τεχνολογικής καινοτομίας, τα όρια στον ανταγωνισμό κτλ. Σε κάθε μία από αυτές τις συζητήσεις πάντα προέκυπτε το θέμα των δεδομένων. Με ένα τέτοιο τρόπο που δεν είχαμε συνειδητοποιήσει και δεν είχαμε αντιμετωπίσει ποτέ στο παρελθόν. Στην πραγματικότητα είναι η ε, ιδιοκτησία ιδιωτικών εταιριών, αλλά που προέρχονται από τη συμπεριφορά ε, των απλών πολιτών. Και γι' αυτό δεν μπορεί να είναι απλώς ιδιωτικά δεδομένα και να τα, εποφελ... να τα εκμεταλλεύονται ιδιωτικές εταιρείες. Αυτά θα πρέπει να αρχίσουμε να τα θεωρούμε ως κοινό αγαθό. Αυτά τα συνολικά, ανώνυμα ε, αγαθά, ας πούμε. Και, είναι και θα πρέπει να είναι και η διοκτησία των α, ε, κρατών μελών. Ε, θα ήθελα να μου πείτε τι άποψη έχετε για αυτό το θέμα, για αυτά τα δεδομένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι πολύ καλή ερώτηση. Θα έρχομαι πιο συχνά γιατί τονίσατε όλες τις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίσουμε. Να απαντήσω ως εξή. Ναι, πρώτα ως στατιστικολόγοι, ναι, μας αρέσει να παίζουμε με τα δεδομένα και να αναζητούμε κάποιες νέες ευκαιρίες. Προσπαθούμε λοιπόν να δούμε με τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες πώς θα χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά τα δεδομένα, τα νέα δεδομένα από τα κινητά συστήματα, από το facebook, το twitter, συνεργαστικές ε, συνεργατικές με συγχωρείτε πλατφόρμες ε, για να τα χρησιμοποιήσουμε στα επίσημα στατιστικά στοιχεία. Και ακριβώς ε, καταλήξαμε στο ότι στις περισσότερες περιπτώσεις τα δεδομένα αυτά μπορούν να συμπληρώνουν τις υφιστάμενες πηγές για να έχουμε παραγωγή στατιστικών στοιχείων αλλά έχουμε μία ας πούμε επαγγελματική συζήτηση. Αυτό το οποίο είναι πιο σημαντικό για το κρατήριο εδώ είναι ότι ενώ κάνουμε αυτήν την έρευνα βλέπουμε κάποια θεμελιώδη προβλήματα. Το πρώτο είναι η πρόσβαση σε αυτές τις πηγές δεδομένων που συνήθως είναι ιδιωτικά δεδομένα. Ε, αυτό είναι ένα θεμελιώδες ζήτημα γιατί για να υπάρχει να υπάρχουν βιώσιμα στατιστικά στοιχεία πρέπει ακριβώς ε, να έχουμε μία ε, σταθερή υπάρχει αυτών των στοιχείων και εδώ πέρα θα μπορούσατε τα επόμενα πέντε χρόνια να παίξετε έναν σημαντικό ρόλο γιατί όπως είπατε είναι ένα θέμα το οποίο αφορά ακριβώς την οικονομία των δεδομένων και ποιος είναι ο ρόλος των δεδομένων στην εφαρμογή της ε, πολιτικής. Και αυτό είναι ένα ερώτημα. Παραδείγματο χάρη ε, οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες ε, όλες ετοίμασαν ένα έγγραφο θέσεων, πάρα πολύ σπάνιο αυτό, να ενωθούν όλα τα κράτη-μέλη και να υπάρχει η πρόοδο στα δεδομένα. Το δεύτερο αφορά ακριβώ την εμπιστευτικότητα και την ιδιωτικότητα των στοιχείων και έχουμε τον κανονισμό που τη τίθεται ισχύει στις 18 Μαΐου και έχουμε κάποια ρεαλιστικά ζητήματα που πρέπει να λυθούν από τις στατιστικές υπηρεσίες γιατί έχουμε χρήση ιδιωτικών δεδομένων ή δεδομένων από ψηφιακές πηγές όπως ε, τα λέμε, τα δεδομένα που δημιουργούν ε, οι μηχανές, υπάρχουν ζητήματα ιδιωτικότητας. Ε, όπως βεβαίως ζητήματα που αφορούν την προστασία των δεδομένων. Οπότε προχωράει η καθαρά στατιστική εργασία, αλλά υπάρχει και το ζήτημα των υποδομών, της πρόσβασης, αν πρέπει να πληρώνουμε για τα δεδομένα, αν πρέπει να είναι ανώνυμα. Και βεβαίω ε, είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι αρκετά περίπλοκο. Σας ευχαριστώ. Ε, διαβάζουμε εντωμεταξύ το τι συνέβη με την χρήση αυτών των δεδομένων από κάποιες άλλες εταιρείες. Και υπάρχει ανησυχία για το θέμα αυτό. Ή πρέπει Το θέμα του προ, προλαλήσαντος ε, του Ιταλού συναδέλφου ε, με φέρνει σε κάτι που θέλω που είπα και εγώ στην αρχή της παρέμβασής μου τα σεξι μεγαλοδεδομένα ε, και πώς ε, παντρεύονται με τις παλιές παραδοσιακές ε, στατιστικές να σταθώ λίγο σε αυτό. Είπατε ότι οι εθνικές αρχές κινητοποιούνται για αυτό το θέμα, τα μεγαλοδεδομένα δηλαδή, τα big data. Έχετε κοινέ συζητήσει, πώς κινητοποιούνται. Κινείστε προς την ίδια κατεύθυνση, είστε στο ίδιο μήκο κύματο σε αυτές τις συζητήσεις. Υπάρχουν εταιρικέ σχέσεις μεταξύ των ε, στατιστικών υπηρεσιών και των παρόχων αυτών των δεδομένων. Και υπό, μία, υπό ποια μορφή θα πρέπει να αλλάξει νομοθεσία, να εξελιχθεί. Μιλήσατε το θέμα της πληρωμής, γιατί είναι από τα θέματα τα οποία ανέφερα και εγώ χθε όταν μιλήσαμε με τον κύριο Τζοβανίνη. Το πρόβλημα του κόστους πρόσβασης σε αυτές τις πληροφορίες. Και βλέπουμε ειδικά στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, η Bloomberg ε, ανέπτυξε ένα μοντέλο ένα μοντέλο πούμε, παρόχου δεδομένων που είναι πανάκριβο ας πούμε και που εξελίσσεται. Γιατί είναι, υπάρχει εκεί κερδοφορία ας πούμε, γι' αυτό βλέπουμε όλο και περισσότερους ε, παρόχους ας πούμε να αντιγράφουν αυτό το μοντέλο, να συλλέγουν πληροφορίες Φαντάζομαι ότι Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες δεν έχουν πρόσβαση εκεί. Πώς μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα αυτή, ε, να την παραβιάσετε. Μπορεί να χρειαζόμαστε αυτές τις στατιστικές. Είναι ένα θέμα, ειδικά για τις χρηματαγορές, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Ε, θα γίνει όλο και πιο σημαντικό αυτό το θέμα. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε όλο και περισσότερες νέες ε, οντότητες, ας πούμε, που συλλέγουν δεδομένα. Τι θα πρέπει να, θα πρέπει να αλλάξει νομοθεσία, θα πρέπει να κάνουμε συμβάσεις, αναπερίπτωση. Πώς θα ε, εντάξουμε και θα λάβουμε υπόψη μας αυτή τη νέα διάσταση. Ε, ε, σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Yes, this is a very important... Είναι πάρα πολύ σημαντική η συζήτηση αυτή και ενδιαφέρουσα. Ναι συνεργαζόμαστε με τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες και μία πτυχή είναι ότι προσπαθούμε να προωθήσουμε την ανταλλαγή απόψεων εκεί όπου έχει αλλάξει η εθνική νομοθεσία για να διασφαλίσουμε την πρόσβαση στα δεδομένα και να υπάρχει συνεργασία. Παραδείγματος χάρη η Γαλλία είναι ένα παράδειγμα που πρόσφατα άλλαξε ο νόμος και είχαμε το πρώτο παράδειγμα για να υπάρχει πρόσβαση σε αυτές τις πηγές. Δεύτερον, έχουμε ακριβώς ε, διαφορετικές ε, συνεργασίες ε, με διαφορετικές συνθέσεις σε συνεργασία με τις εταιρείες κινητής, με την Google, με διαφορετικά δίκτυα, με τα κοινωνικά μέσα και ένα ενδιαφέρον συμπέρασμα είναι ότι και ο ιδιωτικός τομέας τώρα μπαίνει σε αυτήν την διαδικασία και υπάρχει οπωσδήποτε μία ανάγκη για το πώς ε, θα πρέπει να οικοδομηθεί αυτή η συνεργασία. Κάποια στιγμή θα πρέπει να ρυθμιστεί η πρόσβαση στα δεδομένα, στα ιδιωτικά δεδομένα. Ε, το ερώτημα είναι ποιος είναι ο καλύτερος ε, τρόπος ε, να γίνει κάτι τέτοιο. αν θα πρέπει να είναι στον στατιστικό κανονισμό ή σε κάποιους άλλους ε, ειδικότερους ε, κανονισμούς ε. αλλά οπωσδήποτε θα πρέπει να ρυθμιστεί το θέμα. Γιατί οπωσδήποτε δεν υπάρχει κάποια εγγύηση για την σταθερότητα παροχής δεδομένων για στατιστική παραγωγή και χρειάζονται και κάποιοι κανόνες για κάποια σαφήνεια, τι επιτρέπεται, τι δεν επιτρέπεται. Οπωσδήποτε αυτό είναι ένα τομέα που πρέπει να προχωρήσουμε. Σα ευχαριστώ για την διαδικασία αυτή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι σημαντικό κάποιες ε, γυναίκες, με τις γυναίκες μάλλον γενικότερα, να σπάσει η γυάλινη οροφή, όπως ε, χαρακτηριστικά ονομάζεται. Για τα νότατα ε, κλιμάκια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λοιπόν, είναι πολύ καλό που είστε Γενική Διευθύντρια της Eurostat. Και όσα μας είπατε έχουν ιδιαίτερη σημασία. Τα δεδομένα που μας προσφέρετε χρησιμοποιούνται σε πολιτικό επίπεδο και μάλιστα σε περίοδο προεκλογικής εκστρατείας ε, εγώ ως Γαλλικιανή ξέρω ότι αν τα δεδομένα που έχουμε στα χέρια μας όμως ε, τα, θέλει να τα εκμεταλλευτεί κάποιος ε, μπορεί να υπάρξουν πρόβλημα με, τα, με την πολιτική συνοχή λόγω κατά τα διευθυντικά ταμεία. Τώρα, για την ευρύτερη ερμηνεία ενός κριτηρίου. Ως τώρα, στο επίπεδο της πολιτικής συνοχής και σε σχέση με την εδαφική διαχείριση κάποιων ε, κονδυλίων, ε, έχουμε χρησιμοποιήσει μια σειρά από κριτήρια. Όμως, ο αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης, κυρίως το βιωτικό επίπεδο, πολλές φορές κάνει τη χρήση κάποιων κριτηρίων ξεπερασμένη. Η επισφάλεια των θέσεων εργασία, η ποιότητα του επαγγελματικού βίου, η απασχόληση. Αυτά δεν λαμβάνονται πάντοτε επαρκώς υπόψη με τις περιοχές ΝΑΤΣ 3. Λοιπόν, κάποιε περιοχέ εμφανίζονται πλουσιότερε από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Εάν δούμε το βιωτικό επίπεδο όμω δεν είναι πλούσιε. το αντίθετο. Έχουν γίνει πιο επισφαλεί, διότι η ποιότητα τη εργασία είναι κακή, οι συμβάσει εργασία είναι κακέ, οι δημόσιε υπηρεσίε, υπάρχει περισσότερη φτώχεια και ενέργεια και μάλιστα φτώχεια. Μια σειρά λοιπόν από τα κριτήρια που είναι αποτέλεσμα της ε, καθημερινής παρατήρησης της υποβάθμισης της ποιότητας των πολιτών δεν λαμβάνονται υπόψη. Γι' αυτό λοιπόν ως Γενική Διευθύντρια τι μπορείτε να μας πείτε. Η ομάδα μας μπορεί να σας βοηθήσει εάν θέλετε ώστε να χρησιμοποιήσετε νέα κριτήρια διευρυμένη ερμηνεία ε, του πώς θα πρέπει να καταγράφεται το βιωτικό επίπεδο στην Ευρώπη τη στιγμή που παίρνουμε στατιστικά στοιχεία. Η μετανάστευση των νέων. Οι νέοι μας παρατάνε, φεύγουν. Θα λέγαμε ότι είναι περιορισμένοι στο χρόνο, όμως υπάρχει μια τεράστια ομάδα νέων που φεύγουν από ευρωπαϊκά κράτη και πάνε αλλού. Αυτό μειώνει την προσφορά υπηρεσιών, την ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών. Ε, Εάν λοιπόν έχετε σκοπό να διευρύνετε το σύνολο κριτήριο που χρησιμοποιείτε, ευχαρίστω να σα διευκολύνουμε στην Eurostat προσφέροντα σα κάποιε ιδέε για να μελετήσετε και αυτή τη διάσταση. Σας ευχαριστώ. Δώσατε πολλά εμπειρικά παραδείγματα για την σημασία των στατιστικών στοιχείων. Ε, ναι ακριβώς έχουμε τα νέα φαινόμενα, συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη και βεβαίως ε, έχει σημασία να πηγαίνουμε πέρα από τα συγκεντρωτικά στοιχεία, να βλέπουμε μικροδεδομένα την ε, κατανομή τους ε, και βεβαίως να μην αφορά μόνο τις διοικητικές περιφέρειες αλλά και διασυνοριακά τις διαφορετικές ε, κατατάξεις. Δεν είμαστε πια στο θέμα ε, να μην περιοριζόμαστε μόνο στην κατηγορία Δήμου, Επαρχίας, ε, Νομαρχίας κτλ. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και βεβαίως είμαι περήφανη που είμαι η πρώτη γυναίκα γενική διευθύντρια της Eurostat και νομίζω θα έχουμε εμπειρικά δεδομένα ότι μπορούμε να κάνουμε καλή δουλειά. Υπάρχουν τέτοια δεδομένα. Ναι, είμαι σίγουρος, λέει ο Πρόεδρος, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον πολύ ενδιαφέροντα διάλογο. Υπάρχει λοιπόν, βλέπετε, αυξανόμενο ενδιαφέρον ε, για τα στατιστικά στοιχεία και γνωρίζουμε ότι βεβαίως ε, αυτό σημαίνει ότι έχουμε και πάρα πολλά ζητήματα. Και ακριβώς θα πρέπει να συνεχίσουμε τον ε, διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων για να έχουμε και πιο στοχευμένες ε, και συγκεκριμένες ε, εφαρμογές για ε, να τα τυποποιήσουμε όλα αυτά. για να εφαρμόσουμε ακριβώς αυτές τις ρυθμίσεις της συνεργασίας. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ για την προσοχή σας. Ε, πραγματικά ε, δείξαμε ότι είναι πολύ ενδιαφέρον το έργο μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να δώσω την προεδρία τώρα στον Μάρκος Φέρμπερ. Yeah, thank you very much, uh, Roberto. Uh, as we are 10 minutes ahead of schedule, I don't know whether the whole negotiation team was already... Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε 10 λεπτά πριν από το πρόγραμμα. Δεν ξέρω αν έχει φτάσει ο συγητής. μπορεί να περιμένει 10, λίγα λεπτά γιατί δεν έχει έρθει η ομάδα σας. Λοιπόν, ε, διάλειμμα λίγων λεπτών.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

So, colleagues, as uh, we are now in the... Αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε σημείο 12. Πρόταση για κανονισμό Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για την τροποποίηση όσον αφορά την υποχρέωση εκαθάριση, αναστολή υποχρέωση εκαθάριση απαιτήσει αναφορά κλπ. κλπ. Δηλαδή η αναθεώρηση του εμμύρη. Έχουμε λοιπόν το σχέδιο έκθεσης με 32 τροπολογίες. Είχε συζητηθεί τον προηγούμενο μήνα και τώρα έχουμε 135 τροπολογίες. Θα δώσω λοιπόν τον λόγο στον κύριο Λάγκεν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω την ε, γλώσσα μου και επιβεβαιώνω ότι Έχουμε 277 τροπολογίες, ε, οι οποίες ε, όλες σχεδόν ε, πηγαίνουν προς την ίδια κατεύθυνση της μείωσης του κινδύνου και της μείωσης των υποχρεώσεων για τις επιχειρήσεις. Έχουμε λοιπόν τις υποχρέωσεις απαιτήσει αναφοράς ε, για μη χρηματοπιστωτικούς αντισυμβαλωμένους κτλ. Θα τα έχουμε ήδη συζητήσει σήμερα. Το θέμα μας είναι οι τροπολογίες. Θέλω να αναφέρω ακριβώς τον ε, κατάλογο που ε, νομίζω ότι θα απαιτήσει Έχουμε, ε, θα χρειαζόμασταν ίσως περισσότερο χρόνο και έχουμε ακριβώς τον ορισμό του αντισυμβαλωμένου, του μικρού αντισυμβαλωμένου. Εδώ πέρα έχουμε τροπολογίες από διαφορετικές κατευθύνσεις, Σάντερ, Λαμασούν, Χέιζ, Τρεμόζα, Γέτσεκ κτλ. Ε, επίσης όσον αφορά και τον, το, το πεδίο της εφαρμογής και εδώ από την κυρία Σουίνμπερν εδώ θα ήταν δυνατόν ε, στους ορισμούς ε, να καταλήξουμε σε δύο συμβιβασμούς ε, και μπορούμε μετά να διαβουλευτούμε. Έχουμε επίσης και το διμερές αυτό περιθώριο, την αντιστροφή του βάρους της αποδείξεως, δηλαδή αυτοί οι οποίοι θέλουν να ωφεληθούν από την απαλλαγή θα πρέπει να αποδείξουν ότι δεν ξεπερνούν το κατόφλι, οι υπόλοιποι θα πρέπει να συνεχίσουν να κάνουν καθάριση και έχουμε τροπολογίες εμού του κυρίου Λάμπερτς, ε, αντίθετη είναι η κυρία Σουίνμπερν και ο κύριος Φον Βάις Τσέκερ, εδώ έχουμε ένα Ε, πιθανό σημείο διαφωνής. Ε, διαφωνίας. Έχουμε ακριβώς ε, και τον υπολογισμό του ορίου, έχουμε κάποιες μέσες θέσεις πάνω από 30 μέρες μέχρι 12 μήνες και το πώς θα έχει η μέθοδος, δηλαδή αν η Κομισιόν θα εκδώσει μια πράξη κατεξιότηση. Μετά έχουμε την άρση της υποχρέωσης front loading Δεν βλέπω εδώ πέρα κάποια δυνατότητα να δεχτούμε αυτά τα οποία λέει ο κύριος Λάμπερτς ε, και ε, κατόπιν έχουμε τα θέματα των διμερών ε, περιθωρίων και το κατόφλι πάλι για απαλλαγή από την υποχρέωση εκαθάρισης, όλα τα ίδια θέματα. που θα πρέπει να ρυθμιστούν. Μετά έχουμε το λεγόμενο front το Fair, Reasonable, Non-Discriminatory και Transparent, δηλαδή μία πρόσβαση δίκαιη με διαφάνεια χωρίς διακριτική μεταχείριση. Εδώ πέρα συμφωνούν οι περισσότερες ομάδες, η ΕΣΜΑ θα εκδώσει μια οδηγία και θα πρέπει η Κομισιόν και ΕΣΜΑ να εξετάσουν αν θα πρέπει να βελτιωθούν οι αρχές πρόσβασης στην εκαθάριση και το πώς θα μπορέσουμε να αποφύγουμε σύγκρουση συμφερόντων. Και εδώ πέρα έχουμε το άρθρο 4α, το 85 και το εκτιμώντας 9 όπου θα υποβάλουμε κάποιες συμβαστικές προτάσεις. Μετά λοιπόν θα δούμε και το θέμα των ε, αμοιβαίων αυτών κεφαλαίων. Εκεί πέρα προτείνουμε μια πρόταση για τρία έτη από τους κυρίους Βάιτσέκερ, Σουίνμπερν, ε, Φερνάντες κλπ. Για τα δύο χρόνια η κυρία Σουίνμπερν επίσης έχει υποβάλει μια πρόταση παράτασης ε, της εξαίρεσης, ε, μία δηλαδή για διαρκή παράταση δύο ετών. Εδώ πέρα λοιπόν θέλουμε μία συγκεκριμένη έκθεση της Κομισιόν για το εάν είναι πρακτική μια τέτοια λύση εντός δύο ετών από την θέση ενισχύ για να έχουμε επιτέλους μια πρόταση. Μετά έχουμε μια συγκεκριμένη εκθέση της ΕΣΜΑ για το εάν μπορεί να υπάρξει κάποια πρακτική λύση. και βεβαίω ε, σύσταση μια ομάδα συμφερόντων τη Κομισιόν για το θέμα συνταξιωτικών ταμείων. Και εκεί πέρα έχουμε κάποιες μονομένες ε, τροπολογίες των συναδέλφων. Μετά έχουμε την ε, υποχρέωση εκαθάριση όπου έχω τροπολογίες εγώ και ο κύριος Φέρμπερ, αναβολή ενός μηνός, προτείνει ο κύριος Βάιστσέκερ παράταση της ε, απαλλαγής, ε, όχι για παραπάνω από έξι μήνες, εκεί πέρα υπάρχουν διάφορες ε, τροπολογίες. Επίσης θα πρέπει να περιοριστεί το πεδίο εφαρμογής, λένε εδώ πέρα οι κύριοι Λάμπερτς και Σουίνμπερν, εκεί πέρα είναι λίγο δύσκολο να βρεθεί κάποιο συμβασμός. Αναβολή της υποχρέωσης εκαθάρισης σημαίνει και αναβολή της υποχρέωσης ε, trading και εδώ πέρα ε, έχουμε σχετικές τροπολογίες από διάφορα κόμματα και μετά κάποιες μεμονωμένες από τους Σάντερ, Λαμασούρ, Φέρμπερ, ε, Σουίνμπερν, Γέτσεκ και Φον Βάιστσέκα και θα είναι μάλλον δύσκολη η απόφαση. Μετά έχουμε άρση των υποχρεώσεων backloading εδώ πέρα μια τροπολογία λέει ότι η αναφορά των όσων θα γίνουν μέχρι, τις, ε, μέχρι τον 12ο του 2018 είναι υπερβολική επιβάρυνση, εδώ υπό όρους συμφωνώ, για την ιεραρχία των πιστωτών έχουμε και εκεί πέρα τροπολογία, αλλά δεν έχω καταλάβει ε, τι η ιεραρχία ακριβώς ε, προτείνει. Τουλάχιστον είναι κάτι πολύ παρόμοιο με αυτό το οποίο είχα προτείνει και εγώ μετά. Έχουμε το θέμα της ευθύνης ε, στα χρηματιστήρια παράγωγα και τα λοιπά. Δεν θα πρέπει να ε, δούμε μόνο τους κεντρικούς συνοδείς αλλά και τα διάφορα μέρη μας λέει ο κύριος Βαϊστσέκε μετά το αποτέλεσμα της διαβούλευσης ε, και το τι γίνεται με τους ενδο, τις ενδομιλικές ε, συναλλαγές ε, πρώτη να ανακαλύπτονται αυτές παγκοσμίως οι κύριοι Βαϊστσέκερ και λοιποί Χιούμπνερ, Σουίνβερν και τα λοιπά προτείνουν κάτι διαφορετικό ο κύριος Λάμπερτς λέει καμία εξαίρεση εξαίρεση για ενδομιλικές συναλλαγές μόνο όταν ε, και οι δύο εταιρείε ε, είναι στην ίδια κατηγορία, ε, λένε η Σάντερ Λαμασούρ και Βάις Τσέκια. Μετά, οι συναλλαγές over the counter, αναφορά σε μία έδρα, μόνο υπάρχουν διάφορες τροπολογίες, αλλά νομίζω ότι θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε. Ποιότητα των δεδομένων, να αυτό σε πολλά άρθρα και εδώ πέρα θα μπορούσαμε να βρούμε μία λύση σε τέσσερις ε, συμβιβαστικές προτάσεις που δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Μετά έχουμε την επικύρωση των διμερών αυτών περιθωρίων από τις αρχές. Ε, θα πρέπει εντός 12 μηνών να υποβληθεί μία πρόταση για κάποια ρύθμιση με τα FX ε, forwards και swaps στο πλαίσιο των ε, διμερών αυτών κανόνων. Το θέμα είναι τι θα γίνει με τους διεθνείς μετέχοντες στην αγορά. Και εδώ πέρα ακριβώς ε, έχουμε το θέμα της Μεγάλης Βρετανίας και της συγκρισιμότητας εν ώψη του Brexit τα έκθεση αναφορές ε, και αξιολογήσεις για την βελτίωση της διαχείρισης κινδύνου. Και στο τέλος ε, το θέμα phase in ε, και της σταδιακής ισχύως, αν δηλαδή θα τεθεί ισχύ μετά από τρεις ή μετά από έξι μήνες. Συνολικά θεωρώ ότι πέρα από δύο-τρεις ε, επίμαχες ε, τροπολογίες ε, θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε 34-35 συμβιβαστικές και ελπίζω να μην χρειαστεί πάνω από μία συνεδρίαση των σκιωδών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Ισηγητά. Περνάμε στους σκιώδεις. Τον λόγο έχει ο Γιάκουμπ Φον και από του Σοσιαλδημοκράτε. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ κατά πολύ με τον εισηγητή πολλά από όσα έχουμε μπροστά μας είναι πολύ δύσκολο να τα διαχειριστούμε για να βρούμε τις σωστές λύσεις. Μία συνάντηση σκιωδών θα μπορούσε να αρκεί με τον Μπέρν Λάγκεν, αλλά με δύο-τρεις σίγουρα θα τα καταφέρουμε. Είναι ένας τομέας όπου υπάρχει ευρεία συμφωνία και πολύ καλά τα παρουσίασε ο κ. Λάγκεν. Ε, με τα χαρά θα διευκρινίσουμε από κοινού τι ε, πρέπει να αποσαφινιστεί. Σίγουρα θέλουμε την κατάλληλη υποβολή εκθέσεων χωρίς να δημιουργήσουμε υπερβολικό άχθος και ταυτόχρονα να, καθορίσουμε να καθορίσουμε τους σωστούς αριθμούς. Αν κάτι πάει στραβά, η ευθύνη σαφώς πρέπει να αποδίδεται στους αρμόδιους. Να μην καταλήξουμε σε μια κατάσταση όπου στο τέλος κανείς να μην είναι υπεύθυνο αν κάτι πάει στραβά. Είναι και αυτό πολύ σημαντικό για τις συντάξεις. Ένα από τα πιο μεγάλα θέματα εδώ. Απασχολήθηκα με τις ανησυχίες των συναδέλφων και νομίζω το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να σκεφτούμε μακρο, Αλλά είναι και θέμα πολιτικής βούλησης. Θέλουμε να συμβεί ή όχι. Εάν δεν δώσουμε μια όθηση για να προχωρήσουν τα πράγματα, θα χάσει από αυτήν την σωστή καταγραφή ένα μεγάλο μέρο τη αγορά και στο τέλο θα στραφούν πάλι σε εμά και ίσω και εναντίον μα. Εδώ λοιπόν χρειάζεται μια λύση. Δεν είναι πρόβλημα η ήπια και ομαλή μετάβαση. Α δώσουμε μια επιπλέον διετία χρόνο. Αλλά είχαμε και δύο χρόνια για να το σκεφτούμε ούτω ή άλλω. Θα πρέπει λιγάκι να βιαστούμε στην πραγματικότητα και καλό θα ήταν ο χρόνος να είναι περιορισμένος. Να δώσουμε δηλαδή μια όθηση για μια λογική με ένα αλλά και σύντομη στο χρόνο λύση. Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε πώς θα υπολογιστούν και τα ποσά. Είναι σημαντικό για το όλο θέμα του επιλογισμού των περιθωρίων. Για τις αφήσεις αναστολές, κάτι που το έχει εντοπίσει ο Λάγκεν, σε αυτό που ε, βρήκαμε στο, και προτείναμε στην περίπτωση της ανάκτησης και εξυγένσης, εδώ ε, είναι σημαντικό να το ε, ευθυγραμμίσουμε αυτό. Ε, επίσης πρέπει να δούμε αν θα ενσωματωθεί πλήρως αυτό το σύνολο κανόνων. Δεν έχω πρόβλημα. Αλλά εκεί που θα είχα πρόβλημα δεν είναι συνήθω του ομιλού που έχουμε 100% θηγατρική και μια πλήρω ενοποιημένη δομή ομίλου. Τα πράγματα είναι στην πραγματικότητα στην πράξη πολύ περίπλοκα. 60% μετοχέ, α πούμε, και το 40% είναι μοιρασμένο μεταξύ πολλών. οικονομικών και μη οικονομικοί φορεί μέσα σε έναν όμιλο. Να είμαστε λίγο προσεκτικοί, λοιπόν. Να δώσουμε προσοχή και στι λεπτομέρειε όταν σκεφτόμαστε τις συναλλαγές ε, εντός ενός ομίλου ε, για να καταλήξουμε σε μια λογική συμβαστική λύση. Αυτέ ήταν οι βασικέ μου παρατηρήσει και ανυπομονώ για τη συνεργασία μα με τον εισηγητή και του υπόλοιπου κοιόδη για να βρούμε τι κατάλληλε λύσει για την ε, ανατύπωση του ήμυρ. Ευχαριστούμε για του συντηρητικού και μεταρρυθμιστέ και η Swinburne. Ευχαριστώ τον κύριο Λάγκη για την πλήρη του έκθεση που πηγαίνει προ την ίδια κατεύθυνση με τι μου. Ο στόχο τη έκθεσης θα είναι να μην αποδυναμώσουμε το, τη σημερινή δομή ε, όπου οι αναφορές ε, λειτουργούν, αλλά πρέπει να προσαρμοστούν απλώ. Δεύτερο, ο στόχο είναι να μειώσουμε το βάρο του συμμετέχοντε που δεν ε, αποτελούν ε, κίνδυνο για το χρηματοπιστωτικό σύστημα που χρησιμοποιούν ε, ας πούμε τα παράγωγα για hedging. Επίσης θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τα σημερινά κατόφλια, ούτω ώστε να υπάρχει αναλογικότητα για αυτέ τι υποχρεώσει εκαθάριση. Και νομίζω ότι πολλέ από τι τροπολογίε πήγαν προ σωστή κατεύθυνση. Σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογή, ε, για του αντισυμβαλόμενου που δεν ε, πληρούν αυτό το κατόφλι και δεν ε, δημιουργούν πρόβλημα για το χρηματοπιστωτικό σύστημα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ECR θεωρεί ότι μπορούμε να του εξαιρέσουμε από τι υποχρεώσει εκαθάριση. Και μπορεί να είναι μικρά στεξιωτικά ταμεία, μικροί κτηματομεσίτε, Μικρή μη χρηματοπιστωτική αντισυμβαλόμενη λοιπόν. Ε, πρέπει να το δούμε αυτό. Ε, και αν δεν ε, αποτελούν κίνδυνο να μην του εντάξουμε. Σε ό,τι αφορά τα μεγάλα δεξιδοτικά συστήματα, τα οποία λειτουργούν με βάση τι ε, κατευθύνσει ε, για να κάνουν hedging, να κάνουν δηλαδή επιμερισμό του κινδύνου ας πούμε, στι επενδύσει του, πιστεύουμε ότι μια μόνιμη εξαίρεση θα ήταν ε, κατάλληλη. Ε, Όπω λέει και το 254. Πιστεύουμε ότι η αναλογικότητα είναι βασικό στοιχείο. Ε, είναι σημαντικό ε, για την, α, ε, τις υποχρεώσεις αναφοράς. Θα πρέπει να δούμε και τα αποτελέσματα της α, διαβούλευσης για την υποχρέωση αναφοράς και θα πρέπει να δούμε ε, τι καθεστώτα έχουμε για τι υποβολέ εκθέσεων. Πιστεύουμε ε, ότι πρέπει να έχουμε μια συνεκτική προσέγγιση για τη συλλογή δεδομένων, τις αναφορές και την χρήση των δεδομένων. Και αυτή η πρόταση ε, ε, υπάρχει για να μειώσουμε και το άχθος. Το θέλουμε αυτό. Υπάρχει όμως, ε, υπάρχουν και κάποια άλλα επιχειρήματα όπου θα πρέπει να έχουμε μια εξορισμού κατάσταση όπου μικροί ε, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί αλλά και μη χρηματοπιστωτικοί αντισυμβαλόμενοι να μπορούν να βασίζονται στους χρηματοπιστωτικούς αντισυμβαλόμενους για να κάνουν την ε, έκθεση για αυτούς. Ίσως θα πρέπει λοιπόν να ευθυγραμμίσουμε τη γλώσσα για να μην υπάρχει αμφισημία για το ποιος είναι υπεύθυνο ε, γιατί. Και αυτό αφορά και την, ε, τα αποθετήρια ε, συναλλαγών. Ε, δεν νομίζω ότι οι, οι τροπολογίες το αντικατοπτρίζουν. Ε, θα πρέπει να δούμε πολύ προσεκτικά και τις υπόλοιπες, ε, τα υπόλοιπα νομοθετικά κείμενα και να τα ευθυγραμμίσουμε, να ε, υπάρχει μια ευθυγράμμιση με το MIFID και το MIFIR. Μαζί με τον κύριο Λαν και τον κύριο Φέρμπερ θα κάνουμε κοινέ τροπολογίε. Ε, θα πρέπει να δούμε τι υποχρεώσει έχουν ε, η ΜΥΦΙΡ. Ε, θέλει να ταξινομήσει τις εμπορικές συναλλαγές ως μη χρηματοπιστωτικές ε, συναλλαγές. Επίσης υπάρχει ένας ορισμός των ε, swaps ε, με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της Βασιλείας. Ελπίζω συμπληρώνει το, την ιδεολογική σκέψη και λέει ότι θα πρέπει τα swaps θα πρέπει να εξαιρούνται την υποχρέωση ανταλλαγής των περιθωρίων. Ίσως θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα περιθώρια RTS, ε, αλλά θα πρέπει να κάνουμε αυτή τη συζήτηση και να συμφωνήσουμε. Πιστεύω δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Η ε, Επιτροπή αυτή πάντα είχε ισχυρή άποψη για τους μη χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, ε, τις εταιρείες και τη χρήση των παραγόγων. Θα πρέπει να, μπορούν, ε, να μπορεί να γίνει το hedging, να γίνει το επιμερισμό του κινδύνου σε όλες τις δραστηριότητε για τους ομίλους. Δεν θα πρέπει ε, να μπορούν οι ρυθμιστικές αρχές να αποσύρουν την, την άδεια εάν υπάρχει ένας, ε, μία οντότητα του ομίλου ε, που παραβιάζει τους κανόνες. και θα πρέπει να δούμε ποια είναι η πολιτική βούληση. Θέλω να δω τι άλλε τροπολογίε. Ορισμένε ευθυγραμμίζονται με τι δικέ μου τι απόψεις και τι απόψει τη ECR. Πιστεύω λοιπόν ότι ο εισηγητής έχει δίκιο. Θα πρέπει να είμαστε πολύ γρήγοροι ε, και να φτάσουμε σε καλό συμβασμό και καλή ολοκλήρωση. Περιμένω τη συναντήση των σκιωδών και θα συνεργαστώ με όλου του υπόλοιπου ε, σκιώδες εισηγητές. Η φιλελεύθερη Πίτερ Γιάτσεκ από Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως έχω πει και σε προηγούμενες συζητήσεις μας, στηρίζουμε την προσέγγιση του εισηγητή στο συγκεκριμένο θέμα και δεν βλέπω να υπάρχουν σημεία στα οποία υπάρχουν σοβαρές διαφωνίες. Πέραν αυτού όμως μας ανησυχεί η εξαίρεση των συνταξιοδοτικών που ήδη αναφέρθηκε δύο φορές. Είναι σημαντικό για μας να βρούμε μια λύση για να λήξει η περίοδος του νομικού λίμπο της νομικής αβεβαιότητας και γι' αυτό έχουμε υποβάλει τροπολογίες για να διορθωθεί αυτό με την εξαίρεση των συναλλαγών μετά το τέλος της περίοδου εξαίρεσης και την θέση σε ισχύ της, ε, ε, του κανονισμού αναθεώρησης του ΕΜΗΡ. Η Απαλλαγή των χαρτοφυλακίων από τι υποχρεώσει κεντρικού συμβαλωμένου είναι οι μόνε περιπτώσει που θα πρέπει να υπάρχει εξαίρεση για τα αρχεία καταγραφή συναλλαγών, όπω προβλέπει η αναθεώρηση ΕΜΙΡ. Ένα θέμα που δεν έχει θυγεί ω τώρα και όπου δεν έχουν υποβληθεί σχετικώ ανθρωπολογίε, όμω θεωρούμε ότι πρέπει να συζητηθεί μεταξύ των σκιωδών, είναι η έλλειψη σαφήνεια σε ό,τι αφορά την ε, ανάληψη ευθυνών για την ποιότητα δεδομένων σε σχέση με τα αρχεία καταγραφή συναλλαγών. Πρέπει να δούμε πως πρέπει να επιστρέψουμε στη διατύπωση του ε, Μύρ 1 της πρώτης εκδοχής αυτού του κανονισμού όπου ορίζεται ότι είναι η αντισυμβαλόμενη υπεύθυνη για την ποιότητα των δεδομένων. Επίσης για τα θέματα grandfathering. Εκεί θα υποβληθεί μια σειρά από τροπολογίες. Θα πρέπει να δούμε πώς αυτά εφαρμόζονται στα ε, συμβόλαια και τι γίνεται με την αλλαγή της ταξινόμησης. Όσο για το χρονοδιάγραμμα, το διάστημα για την αίσθημα έχει αυξηθεί σε 12 μήνες για να συνάδει και με άλλες προτάσεις νομοθεσίας και τέλος, κατά την άποψή μου είναι σημαντικό, οι συμμετέχοντες στην αγορά να έχουν αρκετό χρόνο για να συντάξουν ε, σωστά τα συμβόλαια βάσει των νέων κανόνων και διατάξεων του ΕΜΗΡ. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει τουλάχιστον ένα τρίμηνο στη διάθεσή τους μετά τη θέση σε ισχύ της πρότασης. Θα πρέπει τα ζητήματα αυτά ε, βεβαίως να τα δούμε και στις κοινέ μας συζητήσεις με τον εισηγητή και τους υπόλοιπους σκιώδες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε με τους πρασίνους. Δεν βλέπω κανέναν. Γκουε. Πάλι δεν βλέπω κανέναν. EFDD. ENF. Η κυρία Κάπελ. Παρακαλώ Μπάρμπαρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι ένα θέμα αυτό στο οποίο υπάρχει μια αρκετά μεγάλη ενότητα όσον αφορά την πρόταση της ε, Κομισιόν και οπωσδήποτε βλέπουμε ότι τα κόστη αναφοράς ε, για τους ε, μη χρηματοπιστωτικούς αντισυμβαλόμενους θα πρέπει να μειωθούν, όπως επίσης και το μήτρο διαφάνειας θα πρέπει να έχει καλύτερη ποιότητα δεδομένων. Αυτά θα τα βάλουμε βεβαίως και στις ε, τροπολογίες μας ε, ότι υπάρχει ακριβώς μια χαλάρωση των προδιαγραφών για τα μέρη της καθάρισης είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό και η εξαίρεση για τα συνταξιοδοτικά ταμεία και οι τρεις αυτές επιλογές ε, όπου θα έχουμε την εξαίρεση αναλόγως με το ποια πρόταση θα είναι επιτάπτους ε, είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό ειδικά για επενδύσεις ε, από πλευράς των συνταξιοδοτικών ταμείων όσον αφορά τις υποχρεώσεις εκαθαρίσεων για μικρούς ε, χρηματοπιστωτικούς ε, παίκτες. Ε, νομίζω ότι και αυτό είναι σωστό. Καλύτερη πρόσβαση στην εκαθάριση και αυτό αναφέρθηκε και να υπάρξει υποχρέωση των υπηρεσιών εκαθάρισης να προσφέρουν δίκαιους όρους ε, είναι νομίζω πάρα πολύ σημαντικό. Θα συνεισφέρει σε βελτίωση και όπως είπε και ο εισηγητής και πολλοί συνάδελφοι χρειάζεται οπωσδήποτε ε, να υπάρξει μια διευκρίνηση για τις υποχρεώσεις αναφοράς, για τις υποχρεώσεις εκαθάρισης, για το κατόφλι εκαθάρισης, για τα ταμεία ακινήτων ε, και εδώ πέρα θα υποστηρίξω την σχετική τροπολογία όπως και αυτό το οποίο είπε ο εισηγητής για την εναρμόνιση των διατάξεων σε σχέση με την εκαθάριση σε ένα παγκόσμιο επίπεδο. Τουλάχιστον να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, δηλαδή να ξέρουμε τουλάχιστον πόσο υψηλά είναι τα ποσά όταν μιλάμε για τα παράγωγα, μιλάμε για ένα ύψος 440 δισεκατομμυρίων ευρώ. Έτσι θα μειωθεί και το κόστος και θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί στην ρύθμιση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Περνάμε λοιπόν στο CatchDI. Μία σύντομη παρατήρηση θα κάνω καθώς έχω ήδη υποβάλει όλες μου τις ε, τροπολογίες. Σας ευχαριστώ γι' αυτό και υπάρχει ακριβώ το θέμα του συγχρονισμού των κανονισμών ΕΜΙΡ και Μύφη είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε, αλλιώς θα έχουμε αυτές ακριβώς τις διαφορές μεταξύ των υποχρεώσεων ε, εμπορίας και εκαθάρισης. Αυτά από μένα ως μια σύντομη παρατηρήση και τώρα έχουμε την Περβάνος Μπερές, παρακαλώ. Ε, ναι. Και εγώ συμμερίζομαι την ανησυχία ακριβώς του σκιώδου συγητή του κυρίου Γιάκο Φάιτσερ. Με τα συνταξιδοτικά ταμεία μπορεί να έχουμε κάποιες αναταραχές. Να δούμε πώς θα τα εντάξουμε στο όλο σύστημα, ιδίω αφού έτσι κι αλλιώς ευθύς εξ αρχής, εάν ε, περάσουμε στο ΕΜΙΡ, την επόμενη γενιά του ΕΜΗΡ ενώ στην ομοθεσία υπάρχει. Σήμερα προφανώς το μοντέλο έχει αλλάξει, αλλά η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί. Η πρόταση του συγγητή να υπάρχει σχέση και διασύνδεση με την πάροδο του χρόνου δεν είναι πολύ ρεαλιστική προσέγγιση του ΕΜΗΡ είναι καθαριστική, είναι refit αυτό που προτείνεται. Αλλά θέλουμε να σταματήσει και το σύστημα αυτών των εξαιρέσεων, εφόσον ε, ε, εντοπίσαμε ότι η αποζημίωση είναι ένας καλός μηχανισμός ακόμη και να διασφαλίσουμε τη σταθερότητα των αγορών. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τις συντάξεις, οι προτάσεις του σκιώδου εισηγητή των σοσιαλιστών είναι και ευστοχές και αρκετά λογικές για να υπάρχει και το κατάλληλο phasing είναι όπως λέμε σε πολύ καλά Βρυξελιώτη. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να φροντίσουμε να ενταχθούν σε αυτό το σύστημα τα συνταξιωτικά ταμεία και να φροντίσουμε να μην ξεφύγει μια ολόκληρη κατηγορία. Τα επιχειρήματα που είναι υπέρ της συμπαράταξης με το ΑΜΙΦ ε, προβλέπουν την εξαίρεση, αλλά όχι εξαίρεση μόνο για αυτήν την περίπτωση, εξαίρεση και για τις ε, συναλλαγές συμπίεσης όπου θα βγει ένα μεγάλο μέρος εκτός αγοράς ή εξαίρεση από τις προϋποθέσεις για την αποζημίωση. Αλλά εδώ μην βρεθούμε με τρύπα στους κανόνες. Η αποζημίωση είναι ένας κανόνας. Θέλουμε να τον εφαρμόσουμε όπου πρέπει. Μην ε, πέσουμε στην παγίδα της, του, της πολλαπλασιασμού των εξαιρέσεων για τις προσωρινές ε, προϋποθέσεις αναστολής επίσης. Εδώ νομίζω για τις γενικές γραμμές και εκεί όπου θα μπορούσαμε να καταγράψουμε τα RTS για τις συνθήκες αποζημίωσης, παρόλα αυτά πρέπει να έχουμε ένα πλαίσιο πολύ σαφές στο πρώτο επίπεδο. Αυτά λοιπόν περιλαμβάνει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καλύπτουν αρκετά τις ανησυχίες των ΜΕΝ και των ΔΕΝ. Thank uh, Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλει η Κομισιόν τον λόγο. Δίνω λοιπόν τον λόγο πάλι στον εισηγητή μας, τον κύριο Λάγκεν. Θα είμαι σύντομος. Ε, τα έχουμε αναφέρει τα διάφορα ζητήματα και τις διάφορες απόψεις ε, και επεξεργαστεί σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, στήριξη όλους. Τώρα εγώ και το γραφείο μου θα επεξεργαστούμε κάποιες συμβιβαστικές προτάσεις και θέλω να υπενθυμίσω αυτό το οποίο είπε τώρα η κυρία Πέρες που προσπάθησα να το παρακολουθήσω όσον αφορά τα συνταξιωτικά ταμεία. Είμαστε πολύ κοντά με τις ε, τροπολογίες. Ε, η γενική κριτική την οποία ασκήσατε δεν υπάρχει ε, αυτό το οποίο λέτε ούτε στις τροπολογίες ούτε κάπου αλλού εγώ το ζήτησα. Νομίζω θα βρούμε κάποιες λογικές συμβιβαστικές ε, λύσεις. Τώρα αν θέλουμε κάποια γενική εξαίρεση όπως ζήτησε η κυρία Έστερ Ντελάγκε αν θέλουμε δύο και τρία χρόνια μετά να έχουμε κάποιες δυνατότητες παράτασης όπως ζητάει η Κομισιόν ή αν πούμε τρία χρόνια με παρατάσεις και μετά καμία εξαίρεση και τέλος. Ή άπαξ δύο χρόνια. Δεν βλέπω λοιπόν τεράστιες διαφορές ε, μεταξύ των όσων λέμε. Είμαι ευέλικτο ε, σε αυτό το θέμα γιατί θεωρώ ότι είναι λάθος μια γενική εξαίρεση αλλά αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν τεχνικά προβλήματα και η Κομισιόν μέχρι στιγμής δεν έχει αναπτύξει κάτι. Και υπάρχει και αυτό το οποίο πρότεινε ο κύριος Τσέκερ. Δεν βλέπω λοιπόν να έχουμε κάποια σοβαρά προβλήματα. Οπωσδήποτε θα βρεθεί ένα συμβιβασμό που θα τους ικανοποιήσει όλους. Εντάξει, Στέρντε Λάγκε θα είναι κατά γιατί έχουν κάποια ε, ιδιαίτερα συμφέροντα οι Ολλανδοί να έχουν τα συνταξιδοτικά του ταμεία εκτό ευρωπαϊκή Εποπτεία. Δεν θα συμπορέσουν να συμφωνήσουν όλοι, αλλά υπάρχει νομίζω μια ξεκάθαρη ε, πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο. Αυτά τα οποία είπε λοιπόν ο Γιάκομπ και ο Πέτερ και ο Μάρκους ε, εκεί πέρα. Θα δούμε τι αποτελέσματα θα έχουμε στο επίπεδο 1 και μήπως θα πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω από πλευράς ε, εκαθάρισης ε, και διευκρινήσεων ε, ή όχι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν. Σας ευχαριστούμε και καλή τύχη στις διαπραγματεύσεις. Ψηφοφορία προβλέπεται σε ένα μήνα περίπου στις 24 Απριλίου. Εάν είστε έτοιμοι και θα πάει στην Ολομέλεια τον Μάιο. Δεν ξέρουμε όμως πότε ακόμα. Εξαρτάται από την ημερήσια μας διάταξη. Ναι, παρακαλώ. Να κάνω μια πρόταση για το χρονοδιάγραμμα. Μέχρι το τέλος της πράσινης εβδομάδας ή στις 9 Απριλίου θα υποβάλουμε τις συμβιβαστικές προτάσεις με την παράκληση να έχουμε κάποια τοποθέτηση και θα πρότεινα ε, να έχουμε την πρώτη συνεδρίαση των σκιωδών συνδυνστών στην, ε, στο Στρασβούργο του Απριλίου. Καλώς. Ωραία. Η διαπραγματευτική ομάδα για το επόμενο θέμα ακόμα δεν έχει έρθει και προβλέπεται να έρθει σε 10 λεπτά και πάλι κάνουμε ένα διάλειμμα λίγων λεπτών.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

Λοιπόν, Πάμε στο σημείο 13 του, της ατζέντας, ε, έλεγχος των άμεσων ξένων επενδύσεων. Ο εισηγητής μας είναι ο Ρόμπερτ Τσίλερ. Τσι... Έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ που με περιμένατε, Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη, συνάδελφοι, που καθυστέρησα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι υποστέριξαν ή υπόβαλαν τι ε, τροπολογίε του στην έκθεση. 105 τροπολογίες έχουμε που δείχνει τη σημασία της νομοδότηση αυτής. Έχουμε πάντα, ω συνήθω, τι πολιτικέ μα διαφορέ. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχει και ομοφωνία. Οι, γεν... οι ξένε επενδύσει θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σοβαρά και θα, ε, και θα πρέπει να τι ελέγχουμε ορισμένε από αυτέ σε ορισμένα κράτη-μέλη. Γι' αυτό μιλάμε για την κρίσιμη τεχνολογία, κρίσιμε υποδομέ. Ε, ε αυτέ οι συμφωνίε θα πρέπει να προστατεύονται. Ε, είμαστε σε φάση συμβιβασμού και χαίρομαι που οι ομάδε συμφωνούν και τα, α, και τα ΜΜΕ είναι κρίσιμη υποδομή. Υπάρχει στήριξη του ορισμού των ε, άμεσων ξένων επενδύσεων από τις πολιτικές ομάδες. Δεν μπορούν να χρησιμοποιούν τα καταχωρημένα αποθετήρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, για να κρύψουν ε, διάφορες επενδύσεις και τους ιδιοκτήτες. Προσπαθούμε να κοιτάξουμε τις τελευταίες λεπτομέρειες ε, γιατί για τα περισσότερα θέματα έχουμε καλούς ε, συμβασμούς. Θέλω στην επόμενη συνάντηση των Σκιωδών να συζητήσουμε το άρθρο 347 για τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου κανένα κράτος μέλος δεν θα είναι υποχρεωμένος να αποκαλύπτει πληροφορίες που είναι αντίθετο προς τα βασικά του συμφέροντα. Το συζητήσαμε εδώ. Ε, ο εισηγητής της ΣΥΝΤΕ ε, και εμείς οργανώσαμε μία ακρόαση για, την, για τον έλεγχο ε, και είχαν και τα κράτη-μέλη εκπροσώπους που είπαν τη δική τους εμπειρία από τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων. Και φτάσαμε στο συμπέρασμα ότι τα περισσότερα κράτη-μέλη καταλαβαίνουν ότι αυτά τα ουσιαστικά συμφέροντα, όπως ασφάλεια, ας πούμε, είναι υπεράνω όλων. Γι' αυτό θα πρέπει να βασιστούμε στη συνθήκη για να βρούμε μια καλή υποσημείωση για αυτό το θέμα. Γενικά προσβλέπω στη συνεργασία για να ρυθμίσουμε τις τελευταίες διαφορές συνάντησης των σκιωδών εισηγητών. Όπως σας είπα, νομίζω ότι πιστεύω ότι θα φτάσουμε σε καλό συμβιβασμό και θα πετύχουμε τη σύνταξη μιας καλής γνωμοδότησης. Οι σκιώδεις εισηγητές από το ΕΛΚ ευχαριστώ, ευχαριστώ τον εισηγητή και το σύνολο των σκιωδών εισηγητών για τη δουλειά που κάνανε ή τη δουλειά που κάναμε μάλλον μαζί. Θέλω να τονίσω την ανάγκη να εφαρμόσουμε αυτό το μηχανισμό και να συντονιστούμε και να οργανωθούμε για να διευκολύνουμε αυτή την ανταλλαγή πληροφοριών. Αυτό το εργαλείο το οποίο θέλουμε να εφαρμόσουμε είναι σημαντικό για να προστατεύσουμε την ε, κυριαρχία μας, για να προστατεύσουμε τις επιχειρήσεις μας και κυρίως αυτές που έχουν, ε, όταν πρόκειται για τις κρίσιμες τεχνολογίες. Δεν θα πρέπει να είναι ένα σύστημα το οποίο θα φοβήσει τους ε, επενδυτές. Νομίζω ότι μπορεί να, φέρει και μια να επιφέρει μια ασφάλεια δικαίου για τους επενδυτές. Και τέλος να υπενθυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι... θα πρέπει να μείνει ανοιχτή, λέει η κυρία Σάντερ. Δεν θέλουμε να κλειστούμε στον εαυτό μας, θέλουμε τις ξένες επενδύσεις για την απασχόληση, για την ανάπτυξή μας. Όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και με τρόπο πολύ ρεαλιστικό. Συνολικά, για τη δουλειά μας υπάρχει συνένεση μεταξύ ημών για να βελτιώσουμε το κείμενο της Κομισιόν και να καλέσουμε τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν αυτό το μηχανισμό screening, ελέγχου, Σήμερα 12 χώρες το κάνουν, αλλά αν είμαστε 28 θα είναι καλύτερα. Να τονίσω κάποια σημεία για τις τροπολογίες που κατέθεσαν τα μέλη της ομάδας μου και που υποστηρίζουμε. Θέλω να τονίσω την αρχή της αμοιβαιότητας καταρχήν. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό αυτή η αρχή για να δικαιολογήσουμε την, τον έλεγχο και μια ιδιαίτερη προσοχή από τις επενδύσεις των άλλων κρατών μελών, να λάβουμε υπόψη μας και τις πρακτικές των άλλων αυτών κρατών μελών απέναντι στις επενδύσεις τις δικές μας. Να υπάρχει αυτή η έννοια της αμοιβαιότητας λοιπόν. Επίσης, θα ήθελα να μιλήσω για τη φύση του επενδυτή. Είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι μπορεί να είναι άμεσα ή έμεσα ελεγχόμενος από μια κυβέρνηση με διάφορους τρόπους. Θα ήθελα να τονίσω την ανάγκη επίσης να προστατεύσουμε τις πληροφορίες που συλλέγονται, γιατί αυτές οι πληροφορίες είναι στρατηγικές. Θα πρέπει οι επενδυτές να έχουν απόλυτη βεβαιότητα ότι οι πληροφορίες τους θα προστατεύονται ειδικά όταν αφορούν εμπορικά μυστικά. Τέλος. Για να προστατευτούν αυτές οι πληροφορίες που συλλέγονται, να επανέλθω καταρχάς στην ιδέα ότι η Κομισιόν θα πρέπει να έρχεται εδώ και να παρουσιάζει μία έκθεση για τη δράση που είχε, δηλαδή τι έλεγχο έκανε μέσα στην χρονιά που πέρασε, ούτω ώστε να έχουμε μια σχέση, έτσι, ένα διάβλο επικοινωνία Κοινοβουλίου κομισιών και η Κομισιόν να ενημερώνει ε, το Κοινοβούλιο με πληροφορίες όχι λεπτομερείς, αλλά συνολικές ας πούμε, για να προστατεύσουμε τις στρατηγικές πληροφορίες και τις ευαίσθητες πληροφορίες. Σας ευχαριστώ λοιπόν και χαίρομαι που θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση που επέρχεται αυτή η συνεργασία. Σας ευχαριστώ. Από τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ. Θέλω να τονίσω τη σημασία των ξένων των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί η επίπτωση των επενδύσεων αυτών στην οικονομία, η μεταφορά της τεχνολογίας, η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, οι καινοτομίες, οι καινοτομίε σε όλου αυτού του τομεί έχουν μεγάλε επιπτώσει. Είναι σημαντικό να συζητήσουμε στην Ευρώπη για την οριοθέτηση, τα όρια αυτών των ε, επενδύσεων. Όλε οι άμεσε ξένε επενδύσει δεν έχουν την ίδια και πάντα θετική επίπτωση. Η πρόταση κανονισμού προβλέπει τη δυνατότητα να κάνουμε έναν έλεγχο για λόγους ασφάλειας και δημόσιας τάξης ε, και να τον κάνει η Κομισιόν, εάν κάποια project ή προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να επηρεαστούν. Με τις ε, τροπολογίες μας προσπαθούμε να ενισχύσουμε τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Χαιρετίζουμε το γεγονός ότι δημιουργούνται σημεία επαφής για τον έλεγχο των ξένων επενδύσεων σε κάθε κράτος μέλος, αλλά νομίζουμε ότι αυτά τα σημεία επαφής θα πρέπει να τα συντονίζει ένα κεντρικό σημείο επαφής που θα βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύουμε ότι πρέπει να δοθεί μια ιδιαίτερη σημασία και προσοχή στις επενδύσεις ε, που προέρχονται από χώρες που υφίστανται κυρώσεις ή που είναι φορολογική παράδειση ε, με βάση τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου του 2017 ή που βρίσκονται στον κατάλογο των μη συνεργαζόμενων δικαιοδοσιών και χωρών ή άλλες χώρες που συνδέονται άμεσα με αυτές τις χώρες οι δικαιοδοσίες. Θα πρέπει επίσης να δώσουμε ε, ιδιαίτερη προσοχή σε τρίτες χώρες που προστατεύουν ε, τις προσόδους ε, από παράνομες ε, δραστηριότητε, από παράνομες οικονομικές δραστηριότητε. Τα παράνομα κέρδη και πρόσοδοι ε, δεν θα πρέπει να βγαίνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς χώρες που δεν συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι άλλο. Εάν ο τελικός δικαιούχος δεν μπορεί να εντοπιστεί, αυτές οι επενδύσει δεν θα έπρεπε να επιτρέπονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε ποιος κάνει μια επένδυση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι παρελθόν έχει αυτή η εταιρεία, ποιος είναι ο τελικός δικαιούχος. Αυτά είναι πολύ σημαντικά στοιχεία, αν τα ξέρουμε. Αυτά ε, θα συνεδριάσουν οι σκιώδεις εισηγητές στη μία μισή ώρα και θα συζητήσουμε περισσότερο τις τροπολογίες. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστούμε. Και ε, τώρα φιλελεύθερη. Βίρινγκ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρία εισηγήτρια. Έχουμε νομίζω με τις ε, τροπολογίες μια καλή βάση για συμβαστικές ε, λύσεις. Έχω κάποιες παρατηρήσεις. Δεν σκοπεύουμε να περιληφθεί εδώ πέρα η αρχή της αμοιβαιότητας. Οποιαδήποτε κίνηση ε, προστατευτισμού θα πρέπει να πηγαίνει προς αυτήν την κατεύθυνση. Δεύτερον, θέλουμε να αποφύγουμε τα κράτη-μέλη να έχουν βέτο για επενδύσεις στην επικράτεια άλλου κράτους μέλους. Επίσης, δεν θέλουμε να αναγκάσουμε τα κράτη-μέλη να ελέγχουν την κάθε επένδυση και ούτε καν την κάθε επένδυση σε στρατηγικό τομέα. Επιπλέον, δεν θέλουμε να φτιάξουμε έναν κατάλογο των μη στρατηγικών τομέων. Οπότε το προνόμιο του ελέγχου παραμένει στα κράτη-μέλη. Αντιθέτως, ο στόχος μας είναι να δούμε εάν είναι αναγκαίος αυτός ο έλεγχος. Και για να γίνει ακριβώς, για να υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει να υπάρξει το λεγόμενο screening. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει το κράτος μέλος να δημιουργήσει, το κάθε κράτος μέλος να δημιουργήσει έναν τέτοιο μηχανισμό. Επίσης, οποιαδήποτε απόρριψη άμεσων ξένων επενδύσεων θα πρέπει να τηρεί τις διεθνείς δεσμεύσεις που έχει αναλάβει το κάθε κράτος μέλος και η Ένωσή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Από τους πράσινους έχουμε τον κύριο Ουρτασούν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να καλωσορίσω τις ε, προσπάθειες ε, της ηγητού να γίνει προσπάθεια κάπως ε, πιο ισορροπημένη και χαιρόμαστε που βλέπουμε και τα μήμια Καλωσορίζουμε και την δημιουργία της μαύρης λίστας. Βλέπουμε όμως ακριβώς ε, ότι υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες οι οποίες θα ήθελα να αναφέρω. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να τονίσω ότι για την ομάδα μας ε, η κρίση του εάν ε, οι άμεσες ξένες επενδύσεις θα επηρεάσουν την δημόσια τάξη θα πρέπει να σχετίζεται με το εάν έχουμε μετατόπιση της παραγωγής ή επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό. Γι' αυτό υπάρχουν τα ζητήματα του άρθρου 4. Επίσης, για τα κρατικά επενδυτικά ταμεία θα πρέπει να προσθεθεί ακριβώς το ότι θα πρέπει να τηρούμε τις αρχές του Σαντιάγο για την διαφάνεια. Δεύτερον, θεωρούμε ότι υπάρχει κάποιο περιθώριο ενός ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να ζητάει τον έλεγχο κάποιων επενδύσεων που αφορούν το κοινοτικό συμφέρον. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει την δυνατότητα να ζητήσει την ενεργοποίηση του σχετικού μηχανισμού για λόγους ασφαλείας ή δημόσιας τάξης. Και τέλος, ε, θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να δείτε τις τροπολογίες μας 162 και 172 για τον συντονισμό των επενδύσεων. Συμφωνούμε με τους στόχους αυτών των προτάσεων, αλλά υπάρχει κίνδυνος ε, διμερούς ελέγχου των επενδύσεων μεταξύ κρατών μελών, κάτι το οποίο θα αποκαλύψει τις ε, διαφορές ισχύω ε, και θα υπονομεύσει την εθνική κυριαρχία. Οπότε θεωρούμε ότι είναι επιθυμητό να προχωρήσουμε με ένα πιο πολυμερές σύστημα, δηλαδή να δημιουργηθεί ένα φορέα με συμμετοχή κράτων μελών και κομισιών που θα είναι αρμόδιο για τον έλεγχο αυτών των επενδύσεων. Έχουμε και άλλε ε, συναντήσεις οπωσδήποτε οι σκιώδεις και θα τα συζητήσουμε αυτά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Την ΚΟΕ δεν βλέπω κάποιον. Για το ΙΝΕΦ. Ε, Μπερνάρ Μονό, όχι ψιάζει. Δεν θα μιλήσετε ούτε εσείς. Μάλιστα, περνάμε στην οφθαλμοφυρία. Κανείς δεν θέλει το λόγο. Δεν ε, βλέπω κάποιον. Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, παρακαλώ. Δύο α, ε, σύντομες ε, παρατηρήσεις. Δύο σχόλια. Πρώτα απ' όλα για την αμοιβαιότητα. θέλουμε να αποστείλουμε το εξής μήνυμα. Εάν το πρόβλημα της αμοιβαιότητας προσθεθεί μεταξύ των κριτηρίων αξιολόγησης, Τέλο πάντων του screening, της σάρωσης, δεν θα έχουμε πρόβλημα μόνο με τις διεθνείς μας υποχρεώσεις, θα στείλουμε μήνυμα προστατευτισμού, αλλά θα γίνουμε στα βρεθούμε σε αντίθεση με τους άλλους δημόσιο, διεθνείς ε, παράγοντες. ποιοι είναι άλλοι που κάνουν screening και ελέγχουν την αμοιβαιότητα του επενδυτή. Το καταλαβαίνετε, είναι ένα βασικό ε, θέμα μένει η αμοιβαιότητα, αλλά δεν είναι αυτό το εργαλείο για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αμοιβαιότητα. Και το άλλο που θέλουμε να πούμε σύντομα για την φορολογία. Καταλαβαίνουμε ότι η φοροδιαφυγή πρέπει να καταπολεμηθεί η αδιαφάνεια των φορολογικών ε, συναλλαγών ή τέλος πάντων το ποιος είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης κάποιων ε, ποσών και συναλλαγών εδώ δεν είναι όμως αυτό το εργαλείο να επιληθούν τα προβλήματα αυτά. Υπάρχει το ε, νομοθέτημα κατά του ξεπλήματος, υπάρχουν και άλλα εργαλεία. Εδώ έχουμε αρθροπιτά και αποκλειστική ρεμοδιότητα. Αν προσθέσουμε και θέματα φορολογίας θα δημιουργήσουμε μια κατάσταση όπου ξαφνικά ε, θα απαιτείται ομοφωνία από τα κράτη-μέλη και αυτό θα οδηγήσει σε θανάτωση της πρότασης. Ατυχές θα ήταν κάτι τέτοιο. Κάποιες φορές ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Αυτό είναι ένα πρώτο βήμα και θέλουμε να συμπαρασύρουμε όσο περισσότερα κάτι μέλη γίνεται. Μην επιβαρύνουμε την πρόταση με πράγματα που μπορεί να είναι μεν λογικά, ένα ενιαίο screening, γιατί σε αυτή τη φάση είναι αδύνατον. Πολιτικός είναι αδύνατον. Δεν υπάρχει αρκετή ευαισθητοποίηση και επίγνωση από τα κρατημέλη. Είναι 16 τα κρατημέλη που δεν έχουν καν screening. Εάν λάβουμε όλες αυτές τις πολιτικές αποφάσεις και τα δεσμεύσουμε, θα τους ε, δυσκολέψουμε. Ας ευαισθητοποιήσουμε και να πετύχουμε περισσότερη διαφάνεια. Είναι ένα πολύ απαραίτητο πρώτο βήμα. Και μετά, σε μια επόμενη αναθεώρηση, πάμε και ένα βήμα παραπέρα. Ευχαριστούμε για αυτές τις παρατηρήσεις. Να μην χάσω την ευκαιρία που είμαι πρόεδρος. Αλλά να πω ότι ελπίζω να μην περιμένουμε τρία χρόνια όπως γίνεται στην εκλογική μου περιφέρεια ξένοι επενδυτέ έχουν επενδύσει στις εταιρείε τη περιοχή και εγώ τώρα πια δεν έχω τη δυνατότητα να αγοράσω καν μια εταιρεία στην Κίνα γιατί οι ξένοι επενδυτέ έχουν ε, καταλάβει το σύμπαν. Τέλος πάντων, η προσωπική παρατήρηση ήταν εκτό ε, διεξαγωγή τη συζήτηση, ο λόγο πάλι στον κύριο Ζήλε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ όλους όσοι μίλησαν εκ μέρου των ομάδων του και την εκπροσώπη τη Επιτροπή και απλώ να πω για το επίπεδο των κρατών μελών. Πολύ σημαντικό αυτό που είπατε. Α ξεκινήσουμε με ένα σύστημα screening σε όλα τα κράτη τη Ευρωπαϊκή Μέλωση και μετά σε όλα τα κράτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά βλέπουμε τι θα γίνει. Πάντω, σε γενικέ γραμμέ, στην ε, Γερμανία υπάρχει ένα σύστημα screening και ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό που ακούσαμε και στην ακρόαση που διεργάνωσε ο κ. Πρόστ στην ε, Γερμανία με του Κινέζου επενδυτέ. Υπήρχε δυνατότητα να υποθεί και να όχι. Αλλά αυτό δεν μπορούσε να γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά στο γερμανικό. Αυτό που ανακαλύψαμε αυτέ τι ακροάσει είναι ότι είναι πολύ διαφορετικά τα συστήματα του screening. Ακόμη και στον Ηνωμένο Βασίλειο, λόγω χάρη, τη Γερμανία ή άλλε χώρε, την Ισπανία που χρησιμοποιούν το screening, τις 12 χώρες που έχουν screening είναι σημαντικό να δούμε τις διαφορές και στην τελευταία συνάντηση των σχεδόν να τα δούμε όλα αυτά από κοινού και με τις υπόλοιπες κοινοβουλευτικές επιτροπές που είναι αρμόδιες για το θέμα αυτό, να καταλήξουμε σε μια καλή συμβαστική λύση πριν την Ολομέλεια. Σε αυτές τις κατευθύνσεις θα κινηθώ. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρο, ευχαριστούμε πολύ. Η ψηφοφορία προβλέπεται για την ερχόμενη εβδομάδα. Ελπίζω λοιπόν να ολοκληρώσετε τότε και η Επιτροπή ΙΝΤΑ που είναι καθήλυνα αρμόδια μάλλον θα ψηφίσει στις 17 Μαΐου και θα δούμε πότε θα περάσει στην Ολομέλεια το θέμα. Είναι προσωρινό το χρονοδιάγραμμα, αλλά η σημαντική ψηφοφορία για μας είναι τις επόμενες εβδομάδες. Ευχαριστώ αυτά για την πρώτη μας συνεδρίαση. Θα σας δούμε το ε, απόγευμα στις 2.30. Λήξεις.